Και πού το γράφει. Πώς ξεκινάει. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σας καλωσορίζω. Θεωρούμε δεκτή την ημερήσια διάταξη σήμερα. Δεν υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Θυμίζω ότι αναμεταδίδεται η συνεδρίαση αυτή από τον δικτυακό τόπο του Κοινοβουλίου. Καλωσορίζω τον ε, Επίτροπο Ντάτσιαν Σόλος που θα μας παρουσιάσει τις νέες προτάσεις για τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με το γάλα και τα προϊόντα τα γαλακτοκομικά. Εδώ και λίγα λεπτά έγινε δεκτή επίσημα η πρόταση αυτή και τώρα διανέμεται, αυτή τη στιγμή διανέμεται η πρόταση. Υπήρχε και η πρόταση για το πακέτο ποιοτικό, ποιότητας μάλλον, αλλά για λόγους εσωτερικής ε, διαδικασίας μόνον αύριο η Επιτροπή μας θα εγκρίνει το λεγόμενο πακέτο για την ποιότητα και θα ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα σε μια επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ τον Ντάτσαν όμως για την παρουσία του. Πρώτα θα δώσω το λόγο στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων να προετοιμαστούν. Θα τους δώσω τον λόγο πρώτους και μετά σε όλους τους συναδέλφους που το επιθυμούν. Ευχαριστώ ε, Επίτροπε. Έχετε το λόγο πρώτος. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως σας υποσχέθηκα στην αρχή του χρόνου, έχουμε πλέον μπροστά σας με μια νομοθετική πρόταση σχετικά με τα γαλακτοκομικά. Έχουμε ζωντανές τις εικόνες της γαλακτοκομικής κρίσης του 2009, όπου οι γαλακτοπαραγωγοί πέρασαν από μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Οι προτάσεις τις οποίες θα σας κάνω σήμερα έχουν σαν στόχο να βγάλουν τα μαθήματα αυτής της κρίσης και να αναλύσουν την κατάσταση στην οποία σήμερα βρισκόμαστε και να χαράξουν τις προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα όπως είπα λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρή κρίση που βιώσαμε πέρυσι, αλλά και τις αποφάσεις για την κατάρ... του Συμβουλίου για την κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων για μετά το 2015. Φτιάξαμε μια ομάδα εργασίας με αντιπροσώπους από τα κράτη-μέλη και από τους επαγγελματικούς εμπλεκόμενους εταίρους και έχουν ε, κάνει κάποιες προτάσεις συστάσεις έτσι ώστε να λάβουμε μέτρα τα οποία θα μας επιτρέψουν να φύγουμε από το σύστημα αυτό των ε, διακανονισμένων ποσοστώσεων <coughs> και ταυτόχρονα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της ανάλυσης που κάναμε της τροφιμικής αλυσίδας γιατί διαπιστώσαμε ότι ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις που γίνονται υπάρχει ένα πρόβλημα σχέσεων εξουσίας ε, και για ορισμένους όπως η γαλακτοπαραγωγή τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ό,τι για άλλους. Στόχος αυτής της πρότασης είναι να διατηρηθεί εν ζωή ο τομέας αυτός, ένας τομέας ο οποίος ίσως ε, αντικατοπτρίζει όσο περισσότερο γίνεται το τι είναι η γεωργία σήμερα. Να καλύψουμε δηλαδή τη ζήτηση και τις αγορές, αλλά να διασφαλίσουμε επίσης και μια κάποια ποιότητα και μια κάποια ισορροπία ε, στην ε, ύπεθρο την ευρωπαϊκή είναι πολύ πιο δύσκολο η γαλακτοτροφία σαν παράδειγμα να μετακινηθεί ή να υπάρξει αλλαγή δραστηριότητας και γι' αυτό ε, εμένουμε στον τομέα αυτό ίσως λίγο περισσότερο. Έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις σχετικά με το τέλος του συστήματος ε, των ε, ποσοστώσεων αλλά θα πρέπει και μετά από το τέλος του συστήματος αυτού, του παρεμβατικού θα έλεγα, να έχουν μια προοπτική η γαλακτοπαραγωγή, η κτηνοτρόφη γενικά. Αυτό είναι απαραίτητο που θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν και θα μπορέσουν να επενδύσουν εκεί που πρέπει και όταν πρέπει, έχοντας τη δυνατότητα δανειοδότησης από τις τράπεζες. Όταν συζητάμε για διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους παραγωγούς και στους καταναλωτές, να θυμίσω ότι τα μέτρα αυτά τα οποία προτείνουμε δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να βάλουν σε χαμηλότερο επίπεδο αυτούς που επεξεργάζονται το προϊόν, αλλά θυμίζω ότι έχουμε άνω των 950.000 γαλακτοπαραγωγών που απέναντί τους έχουν 5.400 ε, που επεξεργάζονται το προϊόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτόν τον συσχετισμό δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Έτσι ώστε όσο περισσότερο γίνεται η παραγωγή αυτή, οι κτηνοτρόφοι, ε, να μπορέσουν να οργανωθούν με σωστό τρόπο και να διαπραγματευτούν με σωστό τρόπο τις τιμές των προϊόντων τους λένε ότι αν αυξηθεί ε, το γάλα θα, στην παραγωγή, στη, στο στάδιο της παραγωγής θα αυξηθεί και σαν τελικό προϊόν που προσφέρεται στον καταναλωτή. Θυμίζω ότι το 2007 όταν ήταν πολύ υψηλό, ε, υψηλή η τιμή του γάλακτος ε, για τον παραγωγό δεν ήταν τόσο υψηλή για τον καταναλωτή. Όταν έπεσε πάρα πολύ για τον παραγωγό το 2009 δεν έπεσε αντίστοιχα. Δεν έπεσε καθόλου ουσιαστικά για τον καταναλωτή η τιμή του γάλακτος. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν ισχύει αυτό που λέγεται ότι επειδή θα υπάρξει μια επανεξισορρόπηση των σχέσεων εξουσίας και του βάρους αν θέλετε που έχουν η παραγωγή από τη μία και αυτή που επεξεργάζεται το προϊόν από την άλλη δεν ισχύει το ότι αυτό θα προκαλέσει αύξηση στην τελική τιμή του προϊόντος στον καταναλωτή. Στόχοι της συγκεκριμένης πρότασης είναι η διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής λειτουργίας της αγοράς. Ειδικό χαρακτηριστικό, ε, η γεωργία παραμένει πάντα ε, μια δραστηριότητα με ειδικά χαρακτηριστικά. Ο προσανατολισμός προς την αγορά, προς τις αγορές και την κάλυψη των αναγκών είναι κάτι το οποίο λειτουργεί αμφίδρομα, δηλαδή πρέπει και οι αγορές να λειτουργούν σωστά έτσι ώστε να μπορέσει και η παραγωγή ταυτόχρονα να λειτουργήσει με ικανοποιητικό τρόπο. Εδώ δεν πρόκειται να επιλέξει κανείς, δεν καλείται κανείς να επιλέξει ανάμεσα στους παραγωγούς από τη μία και στους κανόνες του ανταγωνισμού από την άλλη. Είναι σαφές, ο, σαφής ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους κανόνες για τον ανταγωνισμό στον τομέα της γεωργίας και έχει ξεκαθαριστεί ο τρόπος αυτός και για τον τομέα ε, της παραγωγής γάλακτος. Τι προτάσεις λοιπόν κάνουμε στα πλαίσια αυτού του πακέτου. Καταρχάς θέλουμε να προσφέρουμε την δυνατότητα στον παραγωγό να διαπραγματευτεί συμβάσεις στα πλαίσια των οργανώσεων των παραγωγών με αυτούς που επεξεργάζονται το προϊόν. Προτείνεται η οργάνωση των παραγωγών να μπορεί να δημιουργείται, να συνίσταται ε, στα πλαίσια του 3,5 του συνόλου παραγωγής γάλακτος, χωρίς να ξεπερνά όμως το 33% της εθνικής παραγωγής, το 3,5% σε επίπεδο Ευρώπης, αλλά 33% σε εθνικό επίπεδο. Είπαμε εμείς ότι η πιο σημαντική εταιρεία επεξεργασίας γάλακτος συγκεντρώνει το 3,5 περίπου του συνόλου της γαλακτοπαραγωγής. Και δεν αναφέρομαι εδώ σε συνεταιριστικές οργανώσεις, αναφέρομαι σε ιδιωτικές εταιρείες. Προτείναμε επίσης ένα όριο 33% του εθνικού, της εθνικής παραγωγής, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τον ανταγωνισμό στο εθνικό επίπεδο. Κατελάχιστον τουλάχιστον και να αποφύγουμε την δημιουργία μονοπωλίων και να αποφύγουμε τις καταχρήσεις που θα οδηγήσουν στη δημιουργία μονοπωλίων. Λοιπόν, όλα αυτά σημαίνουν ότι θα υπάρξουν τουλάχιστον τρεις οργανώσεις παραγωγών τουλάχιστον ανακράτος μέλος. Στη Γαλλία υπάρχουν πέντε βέβαια, στη Γερμανία υπάρχουν έξι. Ε, αυτό δικαιολογείται γιατί εκεί οι εθνικές αγορές, οι εσωτερικές αγορές, επειδή είναι οι μεγαλύτερες χώρες της Ένωσης, είναι πολύ μεγάλες και το τεκμηριώνουν. Αλλά παρόλα αυτά είναι κανόνες αυτοί που προτείνουμε, οι οποίοι είναι εύχριστοι για τους παραγωγούς και τους επιτρέπουν να οργανωθούν σωστά και να διαπραγματευτούν καλύτερα τις συμβάσεις τους με αυτούς που επεξεργάζονται το προϊόν, με τις επιχειρήσεις. Αυτές οι συμβάσεις μπορεί να γίνουν ε, ε, υποχρεωτικές στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη όπου, μάλλον εκεί που δεν υπάρχει απόφαση έτσι ώστε οι συμβάσεις αυτές ε, να είναι υποχρεωτικές, οι παραγωγοί μπορούν να διεκδικήσουν την αναγνώριση μιας τέτοιας σύμβασης σαν υποχρεωτική. Δηλαδή δεν υπάρχουν διακρίσει σε βάση περιπτώσει από τη μία χώρα στην άλλη, ανεξάρτητα του αν αναγνωρίζονται οι συμβάσει αυτέ σαν δεσμευτικέ. Εξαιρέσαμε τι συνεταιριστικέ οργανώσει από τον κανονισμό αυτό, διότι διέπονται από ένα ιδιαίτερο οργανωτικό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει και την παραγωγή. Ένα σύστημα το οποίο εμείς δεν θελήσαμε να διαταράξουμε, αλλά εδώ παρενθετικά λέγω ότι τα κίνητρα αυτά τα οποία δίδουμε για την οργάνωση της παραγωγής των παραγωγών θα ενθαρρύνουν μέσω πρόθεσμα των παραγωγών να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αν όχι σε συνεταιριστικό επίπεδο να προχωρήσει σε ομαδοποιήσεις παραγωγών για να βελτιώσει τη διαπραγματευτική του θέση. Νομίζω ότι μακροπρόθεσμα είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο έτσι ώστε να εδρεωθεί η θέση του παραγωγού. Γι' αυτό ακριβώς και προσαρμόζουμε τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου έτσι ώστε να υποστηρίξουμε οικονομικά και να ενθαρρύνουμε χρηματοδοτικά την δημιουργία αυτών των οργανώσεων, ομαδοποιήσεων των παραγωγών είτε υπό τη μορφή συνεταιριστικών οργανώσεων είτε υπό κάποια άλλη μορφή όταν το θελήσουν, όταν το επιθυμήσουν οι παραγωγοί. Έχει τεθεί ένα όριο για τις προτάσεις αυτές χρονικό μέχρι το 2020. Ο κανονισμός αυτός θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το 2020. Χρειάστηκε επίσης να υπάρξει και μία μεταβατική περίοδος για τις προτάσεις αυτές. Προβλέπονται φυσικά και ορισμένες εξαιρέσεις, σύμφωνα πάντα με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ενθαρρύνουμε τον παραγωγό να προχωρήσει σε ένα νέο οργανωτικό σύστημα, σε ένα σύστημα συνεταιριστικό, ε, των παραγωγών. Βάζουμε επίσης και τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να υπάρχουν για το σύνολο της επαγγελματικής δραστηριότητας. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέψει την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών στην τροφιμική αλυσίδα ανάμεσα σε αυτόν που παράγει και σε αυτόν που επεξεργάζεται με τον τρόπο αυτό. Από τη μία ενθαρρύνουμε την υπογραφή συμβάσεων και την διαπραγμάτευση συμβάσεων ανάμεσα στον παραγωγό και αυτόν που επεξεργάζεται και ταυτόχρονα δημιουργούμε το πλαίσιο διαλόγου ανάμεσα στις διαφορετικές αυτές επαγγελματικές κατηγορίες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και δημιουργούνται μορφές συνεργασίας διαφορετικές από αυτές τις οποίες προβλέπουν απλά οι συμβάσεις. Έρευνα, ποιότητα, ανταλλαγή χρηστών πρακτικών Νομίζω ότι εκεί όπου δεν υπάρχουν αυτές οι επαγγελματικές οργανώσεις πρέπει να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία τους και την ανάπτυξή τους. Τα συστήματα αυτά και οι δομές αυτές ισχύουν για ορισμένους τομείς όπως τα οποροκυπευτικά και πήραμε τα καλά παραδείγματα που έχουμε σε κάποιους τέτοιους τομείς όπως τα οποροκυπευτικά για να τα εφαρμόσουμε και στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής. Υπάρχουν επίσης προτάσεις τις οποίες κάνουμε σχετικά με τη διασφάλιση της διαφάνειας ενισχύοντας σε κοινοτικό επίπεδο την εποπτεία των αγορών, της εξέλιξης των τιμών, της εξέλιξης των ποσοτήτων παραγωγής και των προοπτικών γενικότερα, των τάσεων στην κατανάλωση και έτσι συλλέγουμε δεδομένα τα οποία θέτουμε στη διάθεση των εμπλεκομένων στον συγκεκριμένο τομέα για να μπορούν να διαπραγματεύονται τις συμβάσεις τους εν γνώση των λεπτομεριών και των χαρακτηριστικών της συγκυρίας. Και έτσι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα βελτιώσει τις δυνατότητες διάδοσης και κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών στα πλαίσια ενός κάποιου ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου το οποίο θα συγκεντρώνει τους αντιπροσώπους των κρατών μελών αλλά και τους αντιπροσώπους γενικότερα της αλυσίδας παραγωγής έτσι ώστε να είναι συστηματικά διαθέσιμα τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε. Αυτές είναι οι προτάσεις τις οποίες κάνουμε. Τώρα θα έλεγα ότι το παιχνίδι εσείς θα το κάνετε. Εσείς και το Συμβούλιο ελπίζω να μπορέσετε να πάρετε μια κάποια απόφαση το ταχύτερο δυνατόν έτσι ώστε να έχουν στη διάθεσή τους το μέσο αυτό η παραγωγή. Βάλαμε επίσης το όριο του 2020, αλλά βάλαμε και δύο ενδιάμεσες χρονικές, θα έλεγα, στιγμές. Μια πρώτη ανάλυση θα πρέπει να, γίνουμε, να γίνει μέχρι το 2014, το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μια ανάλυση σχετικά το πώς εξελίσσεται ο τομέας μετά την εφαρμογή των μέτρων αυτών, πριν από το τέλος των ποσοστώσεων δηλαδή, και εφόσον είναι απαραίτητο θα προτείνουμε και συμπληρωματικά μέτρα προσαρμογής για την αλλαγή του συστήματος. Και μια άλλη ενδιάμεση ημερομηνία, το 2018, πριν από τον τερματισμό δηλαδή, της περίοδου εφαρμογής αυτού του προτινομένου κανονισμού. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως έλεγε ο Πρόεδρος, η απόφαση ελήφθη επίσημα σήμερα το πρωί, γι' αυτό και σας διανεμήθηκε μόλις τώρα το κείμενο. Αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα είναι μια πρώτη συζήτηση, μια πρώτη επαφή και όταν θελήσετε να κρίνετε μάλλον ότι είναι απαραίτητο, μπορώ να επανέλθω εδώ για να τα συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ λοιπόν τον Επίτροπο. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σου, σε ευχαριστώ για την ταχύτητα με την οποία ήρθες εδώ, αμέσως μόλις έγινε δεκτή η πρόταση αυτή. Ξεκινάμε λοιπόν την συζήτηση. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε λοιπόν δίνοντας το λόγο στους, στους ε, συντονιστές, ιδιαίτερα στον Νίκολσον, ο οποίος θα είναι ο εισηγητής μας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και εφόσον ο Τζέιμς συμφωνεί θα του δώσω πρώτο τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ επίσης τον Επίτροπο που προσήλθε και που μας έδωσε το ε, έντυπο αυτό. Μόλις ε, βγήκε από το πιεστήριο και είναι ένα μικρότερο έγγραφο από τα προηγούμενα που είχαμε στα χέρια μας και είχαμε δει, υποθέτω θα είναι πολύ δύσκολο για μας να κάνουμε μία σε βάθος ε, ανταπόκριση και τοποθέτηση σε αυτό το σημείο. Θα έλεγα ότι είναι έχει δίκιο ο Επίτροπος όταν επισημαίνει τα προβλήματα τα οποία είχαμε σε σχέση με τη βιομηχανία, χαμηλές τιμές και όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζαμε στο παρελθόν. Νομίζω θα πρέπει στην ομάδα υψηλών επαϊόντων να, να ε, ευχαριστήσουμε για την εργασία και για την αξιολόγηση αυτής της πρότασης από την Επιτροπή. Ελπίζουμε ότι πολύ μεγάλο μέρος αυτής της δουλειάς θα έχει ενταχθεί στην τελική αυτή πρόταση της Επιτροπής. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γαλακτοκομικός τομέας, αλλά όχι μόνο αυτός, αλλά και άλλοι πολλοί τομεί στη Γεωργία, είναι το ευμετάβλητο των αγορών και για τη σταθεροποίηση των αγορών ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα είναι θετικό βέβαια. Αλλά επίσης πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι ενώ εμείς στην Ευρώπη έχουμε μείζωνα ρόλο να διαδραματίσουμε για το μέλλον των γαλακτοκομικών, αυτά που συμβαίνουν στην παγκόσμια αγορά έχουν και αυτά τις επιπτώσεις τους. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση μελλοντικά από πλευράς μας. Μία από τις φράσεις που χρησιμοποιούσε ο προηγούμενος όσον αφορά την κατάργηση των ποσοστώσεων ήταν η διασφάλιση της ύπεας προσγείωσης για τον γαλακτοκομικό τομέα και το γάλα. Αυτή θα είναι η πρόκληση που πρέπει εδώ και τώρα εμείς να αντιμετωπίσουμε, να δούμε θα πετύχουμε αυτή την ήπια προσγείωση για τη βιομηχανία, γιατί είναι πολύ σημαντικό πιστεύω η παραγωγή, οι γεωργοί να γνωρίζουν πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον τους και πώς μπορούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο να εργαστούν. Διότι αυτό που χρειάζονται και η γεωργία και η βιομηχανία είναι ένα πολύ σταθερό πλαίσιο για το μέλλον. Σταθερό μέλλον και όχι αβεβαιότητα. Και πρέπει να ξέρουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, πώς θα λειτουργούν οι αγορές και πώς θα δώσουμε συνέχεια σε αυτά και την αξιολόγησή τους. Ως εισηγητής σίγουρα την επόμενη εβδομάδα ελπίζω ότι θα αρχίσω με τις συζητήσεις με άλλους συντονιστές και ε, σκιώδεις εισηγητές στις επαφές μου στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή για να προχωρήσουμε αυτή την έκθεση και να συνεργαστώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέτρο του εφικτού για να διασφαλίσουμε επειδή πιστεύω ότι υπάρχει τεράστια ευθύνη που επομιζόμαστε ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή να διασφαλίσουμε ότι θα καταφέρουμε να προσεγγίσουμε όλα αυτά τα θέματα με ένα ιδιαίτερα λειτουργικό τρόπο, αποτελεσματικό λειτουργικό τρόπο να πετύχουμε ό,τι καλύτερο για τη βιομηχανία και του γεωργού. Προσβλέπω σε αυτό. Ευχαριστώ. Ε, Αρχίσουμε λοιπόν με τους συντονιστές. Έτσι συνήθως κάνουμε. Ο Μισελ Νταντέ έχει το λόγο παρακαλώ. Η κυρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για τον Επίτροπο ο οποίο εφαρμόζει ακόμη για μια φορά το κανόνα για να έρθει να παρουσιάσει εδώ τις προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει από την Κομισιό καθώς επίσης και η απόφαση η οποία λήφθη. Το είπατε προηγουμένως και το είπατε και στην παρουσίασή σας ότι το η παραγωγή εξαρτάται από την αγορά αλλά εξαρτάται και από την έκταση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης ότι η, παραγωγή, γαλακτό παραγωγή είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυσκολία αυτής της εργασίας που είναι από τις πιο δύσκολες μεταξύ των διαφόρων γεωργών της Ευρώπης και αυτό ε, μας κάνει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί σε σχέση με αυτούς, σε σχέση με αυτούς ε, προς αυτούς σε σχέση με τους άλλους. Επιμείνατε πολύ περισσότερο για αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό και η διαπραγματευτική δύναμη η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και έχει αναγνωριστεί μέσα από την κινητοποίηση που έχει γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο των παραγωγών και θα πρέπει να αναλύσουμε αυτή τη στιγμή του αριθμούς που μας δώσατε 3,5 εγώ είπατε 33 σε εθνικό επίπεδο είναι αρκετοί αυτοί οι αριθμοί για να έχουμε ένα βάρος όσον αφορά στην άλλη άκρη. Υπάρχει η μεγάλη οργανισμή διανομή η οποίοι είναι πολύ βαρύς και βαρύνουν στην βλάστηγκα όσον αφορά τη μεταποίηση, με την επεξεργασία, ε, την εργασία η οποία θα κάνουμε, η επεξεργασία των στοιχείων που μας δώσουν που θα κάνουν τις επόμενες εβδομάδες θα μας επιτρέψει να, έχουμε περισσότερο, να ρίξουν περισσότερο φως σε αυτά τα στοιχεία. Επίσης θελήσατε να ενισχύσετε τη διαφάνεια μας φάνηκε σε εμά σαν ΕΛΚ ε, σημείο κλειδί το Άμπερνες το είπε εξάλλου σε μια προηγούμενη αγόρευσή του ότι αυτή η διαφάνεια η οποία θα πρέπει να είναι προς πάντες είναι στο τέλος όλης αυτής της αλυσίδας θα λέγαμε και δεν θα πρέπει να υπάρχει μόνο από την παραγωγή αλλά θα πρέπει να υπάρχει ε, διαφάνεια και στη διανομή του γάλακτος διαφορετικά επανέρχομαι σε αυτό το οποίο είχα πει διότι η διανομή είναι τόσο θα λέγαμε σκοτεινή που δεν διευκολύνει τα πράγματα. Δεν πήρατε εσείς βεβαίως, την, δεν παραλάβατε την ιδέα της ε, καινοτομία. Ήταν μια ιδέα η οποία ε, εξεφράσει εκ μέρους της ομάδας υψηλού επίπεδου. Διαπιστώσατε ωστόσο ότι εάν η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει επενδύσει για την καινοτομία όσον αφορά τα γαλακτοκομικά, η συνεργασία η συνεργασία και οι συνεργατικοί οργανισμοί έχουν ακόμη ανάγκη ένα σπρόξιμο θα λέγαμε αν πραγματικά θελήσουμε να αυξήσουμε και να διαφοροποιήσουμε τη γαλακτοπαραγωγική γαλακτοπαραγωγή συγγνώμη. Βέβαια όλα αυτά δεν θα έχουν αποτέλεσμα εάν δεν καταλήξουμε εντάχει με σπουδή και γιατί μην ξεχνάω ότι αυτό είναι μια πρώτη ύλη γεωργική και μόνο 1% του γάλακτος ήθελε να προσθεθεί το 2009 και βεβαίως οδήγησε αυτό <clears throat> σε μια απορρίθμιση αλλά και την πτώση των τιμών. Μια ερώτηση που θέλω να σας πάω κύριε Επίτροπε μόνο. Το 2008 είχε συμφωνηθεί όπως η Κομισιό να κάνει μία μελέτη όσον αφορά το 2010 και μια άλλη μελέτη για το 2012 ή μήπω έχετε μερικά στοιχεία όσον αφορά αυτή τη μελέτη που έπρεπε να γίνει για το 10 τουλάχιστον γιατί για το 12 είναι πολύ μακριά όσον αφορά πάντοτε σας παραλαμβάνω την αγορά του γάλακτος πανευρωπαϊκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λαμπρά λέει ο πρόεδρος. Ο Μάρκ Ταραμπέλα έχει παρακαλώ το λόγο των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, προφανώς η ανακοίνωση τους ήταν αναμενόμενη, διότι η αγορά του γάλακτος είναι, περνάει μια κρίση που δεν έχει επιληθεί. Και σας είναι βέβαια σχηρότερη από αυτή που υπήρχε πέρσι. Βεβαίως φάλετε σε ένα πλαίσιο αυτό το θέμα και αληθεύει πραγματικά γιατί σαν τον μίλησε είπατε πραγματικά ότι αυτή τη στιγμή είτε το γάλα είτε οι άλλοι τομεί είναι σε, μια, σε έναν αυρασμό και αυτό βεβαίως είναι ο χειρότερος εχθρός. Και η τιμή πέρασε από 45 λεπτά σε 18 λεπτά για το γάλα. Αλλά ο συνάδελφος προλαλή σας είπε ότι στην παγκόσμια αγορά ε, αυτή δημιούργησε την κρίση του 2009 και είναι μόνο 6% του παραγόμενου γάλακτό στον κόσμο. Αυτό το 6% καθορίζει την τιμή και αυτό κυκλοφορεί και καθορίζει την παγκόσμια τιμή επαναλαμβάνω του γάλακτος. Ε, μου φαίνεται παράλογο αυτό το πράγμα διότι αυτό γίνεται πάνω από την εΕ και βεβαίω είναι η Ρωσία αυτή η οποία καθορίζει και θα πρέπει να έχει, να κάνει και αυτή αλλά και εμείς είτε να μιλήσουμε, είτε να μειώσουμε, είτε να απαγορεύσουμε την είσοδο γεωργικών προϊόντων, διατροφικών προϊόντων. Βέβαια, ποιο είναι υπεύθυνο, το Συμβούλιο αποφάσισε, όπω ξέρετε, για το 2005 να καταργήσει τις ποσοστώσεις χωρίς να το υποκαταστήσει από άλλο σύστημα το οποίο προβλεπόταν για να μπορέσει να υπάρξει μια ισορροπία στην αγορά πώς λοιπόν θα ρυθμιστεί αυτή τη στιγμή η αγορά χωρίς βεβαίως να υποθέσουμε ότι θα υπάρχει μια κρίση την οποία γνωρίσαμε πριν δύο χρόνια και μπορούμε να λυπηθούμε πραγματικά ότι αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο δεν έπαιξε το ρόλο που θα έπρεπε να παίξει αυτό το δάμα και βεβαίως με μια αύξηση που θα πρέπει να γίνεται 1% ετησίως στην αύξηση παραγωγής. Κάντε προτάσεις λοιπόν όσον αφορά τις παραγωγούς τις οργανώσεις του στο γεγονό αυτή τη στιγμή δομούνται όλο και περισσότερο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το υπογραμμίσατε και μιλήσατε για τους συνεταιρισμούς. Παίρνω το παράδειγμα του Βελγίου. Το 70% του Βελγίου πηγαίνει σε τρεις συνεταιρισμού γάλακτος. Και είναι ένα σύστημα το οποίο δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε βεβαίω, που έχει όμως το υπέρ, το συν, αν θέλετε, όπως και άλλοι τομείς, στον αγροτικό, φρούτα, λαχανικά κλπ. Είναι όμως ένα σύστημα το οποίο ενδιαφέρον καθότι επιτρέπει τους μετασχηματιστές ή αυτούς που επεξεργάζονται ή αυτοί που καθορίζουν τις τιμές αυτοί οι εταιρισμοί είναι από παραγωγούς, αποτελούν από παραγωγούς και οι οποίοι δεν θα πρέπει βέβαια να τους θέσουμε σε αμφιβολία, να μην τους διαλύσουμε, να μην τους ανισορροπήσουμε η διαπαγγελματική δομή είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο μεταξύ των παραγόντων, παραγωγών, διανομέων, επεξεργαστών κλπ. Το ελβετικό παράδειγμα μου φαίνεται, μας έδειξε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα όριο και σε αυτό το θέμα. Μπορούμε να εμπνευστούμε αυτό το πράγμα και να κάνουμε έτσι ώστε είναι ευκτές αυτές οι δύο επαγγελματικέ οργανώσεις και βεβαίως είναι και αποτελεσματικέ. Μιλήσατε επίσης για τη διαφάνεια, με την παρατήρηση είπατε, παρατήρηση της διαφάνειας. Πιστεύω πως ε, η παρατήρηση δεν θα είναι για την παρατήρηση, αλλά ότι για της παρατηρήσεως θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα παρατηρητήριο των τιμών και των ορίων των τιμών, ούτως ώστε να καθορίζεται πολύ καλύτερη τιμή και να μην έχουμε αυτά τα οποία πράγματα, αυτά τα οποία μας ανησυχούν σε αυτό το ντοσχέ αυτή τη στιγμή. Και μια πρόταση την οποία θα μπορούσα να κάνω εγώ και ίσως στην οποία δεν αναφερθήκατε δεχομένω, διότι δουλεύουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτού, είναι να επεξεργαστούμε εκ νέου για την προώθηση των γαλακτοκομικών ε, προϊόντων. Γιατί μειώθηκε στα παιδιά. Γιατί οι διαφημίσεις για τις σόδες, για τα γαζόζες κλπ. είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες, είναι πολύ πιο δελεαστικές και υπάρχουν ψευτοιατροί οι οποίοι βγαίνουν στη τηλεόραση και λένε τα α και τα β και λένε ότι τα γαλακτοκοπικά προϊόντα είναι κακά για την υγεία και ούτω καθεξής. Νομίζω πως πραγματικά θα πρέπει να γίνει μια προώθηση Μπορεί μια προσπάθεια να γίνει στις καντίνες, στα σχολικές, στα σχολικά κτίρια κλπ. Και νομίζω πραγματικά πως πρέπει να δοθεί μια περαιτέρω όθηση όσον αφορά την κατανάλωση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών ε, προϊόντων. Και νομίζω πως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει, διότι μιλάμε μερικές φορές για τη ρύθμιση της αγοράς, αλλά περάσαμε κρίσεις, περάσαμε και στις κρίση, στην κρίση βλέπουμε ότι η κρίση δημιούργησε τη μείωση εν μέρη της κατανάλωση των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ωστόσο, μπορούμε να επεξεργαστούμε εκ νέου και να βρούμε μια λύση η οποία θα είναι εφικτή και να γνωρίσουμε την έξοδο από την κρίση. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε πίτροπε. Είμαστε εδώ στη διάθεσή σας να συνεργαστούμε, να βελτιώσουμε τη θέση ευελπιστώντας πως το τέλος θα έχουμε φως στην άκρη του της σύραγγας και ιδιαίτερα που θα βοηθήσουν τους παραγωγούς και ιδιαίτερα τους παραγωγούς γάλακτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Μάρκ. George Lyon έχει το λόγο παρακαλώ. Ο George. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Τσόλα, με ιδιαίτερη χαρά σας έχουμε ενώπιόν μας στην δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το έγγραφο το οποίο μας παρουσιάσατε. Παρότι ήταν διαθέσιμο το τελευταίο λεπτό. Βλέποντας τι προστοκούσαμε και τι έχουμε μπροστά μας, σωστά είπατε ότι υπάρχει κάποια επίπτωση από τους ε, αρμόδιους ε, του τμήματος ανταγωνισμού και υπάρχει κάποια μικρή μείωση όσον αφορά το μερίδιο της αγοράς σε σχέση με ενώσεις παραγωγών, σε σχέση με τις αγορές σε εθνικό επίπεδο. Ίσως μπορείτε να επεξηγήσετε αν αυτό θα περιορίσει ίσως ε, τις εξουσίες ή τις δυνατότητες που μπορούν να αποκομιστούν από αυτή την πρόταση. Ταυτόχρονα ενώ μεσα τιμές των ε, γαλακτοκομικών έχουν ε, αλλάξει, πιέζονται και πάλι οι παραγωγοί μας ε, εκ νέου έχουμε ε, μια, ένα πόλεμο γαλακτοκομικών τιμών όσον αφορά το λιανικό εμπόριο. Βλέπουμε μείωση 25% όσον αφορά τις τιμές αυτών των προϊόντων για τους παραγωγούς και σε σχέση με τις τιμές ε, ε, στις υπεραγορές ενώ η βιομηχανία των γαλακτοκομικών δεν είναι στην κατάσταση που βρισκόταν το 2008-2009 δεν υπάρχουν αμφιβολίες ε, για μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και αντιμετωπίζονται σήμερα μέσα στην συμπίεση αυτής ε, της διαμόρφωσης των τιμών. Η αποτίμηση που πρέπει να κάνουμε εμεί ω μέλη αυτή τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή, προσπαθώντα να αξιολογήσουμε τι προτάσει σα, είναι ποια διαφορά θα υπάρξει σε σχέση με του γαλακτοκομικούς, ε, του παραγωγού γαλακτοκομικών επιτόπου. Θα βοηθήσουν αυτέ οι προτάσει κατά κάποιο τρόπο αυτού του ανθρώπου. Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε πιστεύω είναι θα υπάρχει δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες διαπραγμάτευσης ε, σε σχέση με τα προϊόντα τους όσον αφορά τις, ε, την ε, διάθεση στην αγορά όταν βλέπουμε ότι έχει οξυνθεί ο πόλεμος και η αντιπαράθεση αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που πρέπει να ερωτήσουμε και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Εδώ θα ήθελα να μας επεξηγήσετε κάτι, να μας πείτε πώς θα μπορούσε να υποφελήσει αυτό τους παραγωγούς. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο αναφύεται σε όλες τις συζητήσεις με τους παραγωγούς είναι οι σκληρές πρακτικές που αντιμετωπίζουν όταν έρχεται η ώρα να διαπραγματευτούν και να υπογράψουν και να συνάψουν συμβάσεις και συμβόλαια με τις πολυεθνικές μεγάλες εταιρείε. Και εδώ πάλι το ερώτημα που πρέπει να διατυπώσουμε και να απαντήσουμε είναι τα μέτρα εδώ και σε σχέση με τις ε, συμβάσεις ε, θα ε, απαμβλύνουν κάπως ισομές πρακτικές και επιπλέον θα μπορούσατε να επεξηγήσετε γιατί δεν υπάρχει κάποια αναφορά σε σχέση με τη διαμεσολάβηση ή ένα σώμα επιδιατησίας όπως έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να υπάρξει δυνατότητα μιας διαμεσολάβησης όσον αφορά την διαπραγματεύση τέτοιων συμβολέων και συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και ε, εταιριών διάθεσης στην αγορά. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε γιατί αυτό δεν καλύπτεται εδώ. Μήπως ε, η απάντηση θα μπορούσε να ήταν ε, ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο ή στο εθνικό επίπεδο με κάποιο διαμεσολαβητή, κάποια εθνική οργάνωση που θα είχε τέτοιες αρμοδιότητες ώστε να μπορούν να απαμβλύνονται αυτές οι πρακτικές έντονες και ομές πρακτικές σε σχέση με αυτές τις συμβάσεις. Το τρίτο τώρα ερώτημα είναι θα δώσει αυτό μεγαλύτερη σταθερότητα σε σχέση με τον ευμετάβλητο χαρακτήρα των αγορών, θα βοηθήσει να υπάρξει ένα πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο, ένας χρονορίζοντας πιο μακροπρόθεσμος, ώστε να υπάρχει μια, ένα βιώσιμο μέλλον για τους ε, παραγωγούς μέσα σε ένα σταθερότερο πλαίσιο. Νομίζω το τελικό τελευταίο ερώτημα που θα είχα εγώ να διατυπώσω είναι προερχόμενος από τη δική μου χώρα, μια μικρή χώρα που εξάγει παντού προς τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, βλέποντας τώρα εδώ την ε, ε, ομοιότητα ή την παράλληλη τροχιά σε σχέση με τα προκυπευτικά υπάρχει μια ανησυχία για μικρές εξαγωγές σε χώρες ότι θα καταλήγαμε σε μια κατάσταση ιδιωτικών μονοπωλίων σε σχέση με την επανεθνικοποίηση αγορών. Μπορείτε να μας διασφαλίσετε ότι οι κανόνες που θα υποβάλλετε θα αποκλείουν κάτι τέτοιο διότι δεν θέλουμε να υπάρξει με κανένα τρόπο στρέβλωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και όχι να την υπονομεύσουμε. Μπορείτε να μας δώσετε τέτοιε διασφαλίσεις. Ευχαριστώ. Grazie Giorgio, adesso κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και στο Κοινοβούλιο παρουσιάζεται αυτό το, αυτή την πρόταση. Ήταν ένα μεγάλο βήμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σίγουρα αυτό, αλλά και για τους παραγωγούς γρακτοκομικών ήταν ένα πολύ μικρό βήμα, πρέπει να πω. Και νομίζω ότι δεν τα καταφέραμε καλά σε σχέση με τους κανονισμούς ε, που ε, έχουν τώρα συγκροτηθεί. Αν 3-3,5% μπορούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τις ποσοστώσεις ε, να, καθοριστούν. Δεν ανταποκρίνεται αυτό στις πραγματικότητες αγοράς. Στην Γερμανία έχουμε μια κατάσταση μια εταιρεία που 5% συνενώνει Τη Ευρωπαϊκή παραγωγής. Βλέπετε ότι οι προτάσεις σας λοιπόν δεν επαρκούν και στη Δανία επιπλέον που έχουμε μια μεγάλη αρμεκτική βιομηχανία, γαλακτοκομική βιομηχανία που 80% της ε, παραγωγής ε, στο εθνικό επίπεδο διασφαλίζει. Πρέπει να διαρωτηθούμε, αυτές οι προτάσεις σας επαρκούν λοιπόν πραγματικά, δεδομένης τη πραγματικότητα. και επιπλέον σε σχέση με τον αρμόδιο για τον ανταγωνισμό επίτροπο. Δεν ξέρω, μπορούν όλα αυτά να είναι εύληπτα και κατανοητά. Δεν θα πρέπει εδώ να υπάρξει δυνατότητα μεγαλύτερων εξουσιών σε σχέση με τους παραγωγούς ώστε να εξισορροπηθεί η κατάσταση στις αγορές. Μετά είπατε ότι το θέμα της διαφάνειας θέλετε να το επανεγγράψετε στην ημερήσια διάταξη και να έχει σημα... σπουδαιότητα. Απόλυτα σωστό αυτό. Και ανταποκρίνεται και σε αυτά που σε πολλά σημεία εμεί είχαμε διεκδικήσει και απαιτήσει. Ποιε όμω είναι οι συνέπειε που θα συναχθούν στο τέλο επιτήρηση εποπτεία τη αγοράς είναι ένα τμήμα, ένα σκέλος. Αλλά πρέπει να μπορούμε να επέμβουμε, να παρέμβουμε όταν έχουμε και την ε, ε, διάθεση των προϊόντων στην αγορά και βλέπουμε τις μεγάλες αλυσίδες ε, διοχέτευση διάθεση προϊόντων στην αγορά. Βλέπουμε ότι ε, τις αυξήσεις τιμών τις μετακυλίουν στους καταναλωτές και δεν υποφελούνται οι παραγωγοί και αυτό οδηγεί σε ε, διακυμάνσεις. Πώς θα αντιδράσουμε σε σχέση με αυτό το πλέγμα, διότι ε, δεν είναι υπό απόλυτο έλεγχο και η εξουσία των μεγάλων αλυσίδων διάθεσης προϊόντων είναι ακόμα μεγαλύτερη από ότι η εξουσία των μεγάλων γαλακτοκομικών εταιριών. Και βλέπουμε ότι η παραγωγή σε σχέση με το ε, τη σημασία που είχαν και έχουν βρίσκονται σε μη αντίστοιχη θέση όσον αφορά τα προϊόντα τους και τα ωφέλη που θα έπρεπε να μπορούν να αποκομίσουν από αυτά. Πρέπει να υπάρχει μια σαφή προοπτική για του ε, παραγωγού σε αυτόν τον τομέα, έτσι δεν είναι. Και με αυτέ τι προτάσει, και ήδη τότε το είχαμε πει για τα αποτελέσματα τη ομάδα υψηλών επαϊόντων, δεν διασφαλίζεται, πιστεύουμε, ότι οι γεωργοί και οι γαλακτοπαραγωγοί θα έχουν ένα διασφαλισμένο μέλλον. Πρέπει το θέμα των κανόνων τη αγορά και των ποσοστώσεων τη ε, αγορά και των περιορισμών ποσοστώσεων να το ελέγξουμε καλύτερα. Με εκπλήσει κάπω ότι από το παράδειγμα τη Ελβετίας δεν συνάγονται κανόνε για την εξέλιξη και τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών γαλακτοκομικών αγορών. Είναι μια σχετικά μικρή και εύκολα εποπτεύσιμη κατάσταση, η κατάσταση της Ελβετίας και βλέπουμε σε σχέση με την προ... τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί εκεί απέτυχαν και επανέρχονται σε ένα ε, σύστημα που ε, θα εμπεριέχει ε, περιορισμούς ποσοστώσεων και θα αναλάβουν μεγαλύτερη εξουσία και αρμοδιότητες η παραγωγή. Γιατί να μην μεταφέρουμε κάποια τέτοια εμπειρία στο ευρωπαϊκό πρότυπο βλέποντας τι κάνει η Ελβετία. Πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε τις συζητήσεις. Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή μας είχα εκφράσει την πεποίθηση ότι κομματικά θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει η προθυμία και πρέπει να υπάρχει η προθυμία να καταλήξουμε σε συμφωνίες για να συζητήσουμε και τις ποσοστώσεις. Διαφορετικά κάνουμε ένα πείραμα το οποίο μπορεί να αποτύχει σε σχέση με την αγορά. Θα έλπιζα ότι αυτή την πρόταση ως ένα πρώτο βήμα πρέπει να την δούμε που στοχεύει στην ορθή κατεύθυνση αλλά δεν πάει αρκετά μακριά και δεν επαρκεί πλήρω και πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει να ακολουθηθεί αυτό το πρώτο βήμα από άλλα περαιτέρω βήματα ώστε στο τέλος να μπορούμε να πούμε πούμε ότι για τους γαλακτοπαραγωγούς θα υπάρχει ένα διασφαλισμένο μέλλον ως προοπτική γιατί διαφορετικά δεν θα τα καταφέρουμε. Και μετά την κρίση, όπως και πριν από την κρίση, οι αγορές γαλακτοκομικών κάθε άλλο παρά διασφαλισμένο το μέλλον τους έχουν. Υπάρχει αβεβαιότητα και πρέπει να επαναλάβουμε αυτά τα οποία είπαμε στο παρελθόν, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Κλείνω με τους συντονιστές δίνοντας τον λόγο στον Φοντάνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την παρουσία του και τη διαθεσιμότητα την οποία επιδεικνύει. Μας επιτρέπει να είμαστε πρώτοι να... που μαθαίνουμε τα στοιχεία τα οποία μας ε, μετέφερε. Νομίζω ότι όταν ξεκινήσαμε την κοινοβουλευτική μας εντολή εδώ βιώσαμε και μία από τις σοβαρές κρίσεις στην Γεωργία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πράγματα βελτιώθηκαν λίγο και μπορεί να πει κανείς ότι έγιναν καλές προσπάθειες και θα πρέπει οι κανόνες οι οποίοι προτείνονται τώρα να αποβούν και αυτοί θετικοί για τους παραγωγούς μας. Σίγουρα είναι χρήσιμη η οργάνωση των παραγωγών, μια οργάνωση η οποία να έχει ισχυρότερες διαπραγματευτικές ικανότητες και αντιπροσωπευτικότητα. Είναι το θεμέλιο θα έλεγα πάνω στο οποίο θα βασιστούν οι παραγωγοί μας για να υπάρξουν σε αυτήν την δύσκολη αγορά. Θα ήθελα όμως να προσθέσω εδώ ότι η πρόταση η οποία γίνεται να αντιγράψουμε δηλαδή την μέθοδο στα οποροκυπευτικά στη συγκεκριμένη περίπτωση στον γαλακτοκομικό τομέα είναι κάτι μεν το θετικό, αλλά θα συνδέσω το θέμα εδώ και με τις ε, διεθνείς αγορές. Υπήρξε μια κρίση στις τιμές, η οποία όμως ξεκίνησε από την διεθνή αγορά στην οποία εμείς συμμετέχουμε, είμαστε τμήμα της αγοράς αυτής, η οποία είναι απορριθμισμένη και δημιουργεί αυτή την συνεχή απρόβλεπτη κινητικότητα. Και γι' αυτό ακριβώς διαρωτώ με αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κάνει κάτι εδώ. Το θέμα δεν αφορά θα έλεγα μόνο τα γαλακτοκομικά αλλά το σύνολο των γεωργικών προϊόντων. Βλέπουμε ότι κυριαρχούν στις διεθνείς αγορές προϊόντα τα οποία δεν έχουν την ποιότητα των δικών μας. Εμείς φροντίζουμε τους καταναλωτές μας και καλά κάνουμε ελέγχοντας φυσικά και το κόστος ή υποστηρίζοντας τους παραγωγούς για να παράγουν ικανοποιητικά ποιοτικά προϊόντα. Παρ' όλα αυτά η παρουσία μας στις διεθνείς αγορές είναι προϋπόθεση για να εξακολουθήσουν οι παραγωγοί μας να επιβιώνουν. Είδα και τους αριθμούς οι οποίοι δίδονται για το 3,5 του ευρωπαϊκού ε, συνόλου ή το 33% του εθνικού συνόλου θα δούμε αν αυτοί οι αριθμοί είναι οι καλύτεροι. Δεν έχουμε ε, δυνατότητες μαγικές για να ξέρουμε αν είναι σωστά τα ποσοστά αυτά για να αποφύγουμε αυτά τα οποία περάσαμε πέρυσι. Ευχαριστώ τον Φοντάνα και θα δώσω αμέσως το λόγο στον Επίτροπο Τσιόλος έτσι ώστε να υπάρξει μία απάντηση ε, στους συντονιστές και μετά θα δώσω το λόγο και σε άλλους συναδέλφους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. κύριος Νίκολσον, επιτρέψτε να σας πω το εξής. Βεβαίως, είμαι έτοιμος να εργαστώ με σας και τις υπηρεσίες σας ως εισηγητής για αυτή την υπόθεση και να σας δώσω όλες τις πληροφορίες εκείνες και όλες τις λεπτομέρειες. Το κείμενο γραφτεί μόλις σήμερα και δεν υπήρχε να, τη δυνατότητα να έχω περισσότερες ε, λεπτομέρειες αλλά είμαι στη διάθεσή σας για να κάνω το, κείμενο, το επόμενο κείμενο σε επόμενες εβδομάδες. Όσον αφορά τη διαφάνεια, για να φτάσουμε μέχρι το τέλος της αλυσίδα, σε αυτό το σημείο μιλήσαμε για τη διαφάνεια η οποία επιτρέπει τους παραγωγούς και τους ε, τους επεξεργαζόμενους να εργαστούμε γνωρίζοντα τα πράγματα διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται οι διαπραγματεύσει για παράδειγμα και οι συμφωνίες οι οποίες γίνονται και οι συμβάσεις οι οποίες γίνονται η διαφάνεια, το διαπαγγελματικό είναι συνδεδεμένα. Το ένα δεν αρκεί εάν δεν υπάρχουν και τα άλλα. Διότι είναι μια σύμβαση, αλλά δεν υπάρχει ένα πλαίσιο για να μπορεί να υπάρξει αυτό ο γύρος αυτής της όλης υπόθεσης. Το, το πρόβλημα δεν λύνεται. Ο Τζόρτζο Λάιον μίλησε για τον μεσολαβητή. Για μεσολαβητή. Δεν μπήκαμε σε αυτή την λεπτομέρεια γιατί αποφασίσαμε ότι η σύμβαση έχει ένα νομικό υπόβαθρο υπάρχει μια δικαιοδοσύνη η οποία μπορεί να κρίνει αν πραγματικά δεν αρμόζει κάτι. Μήπως θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω από τη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα και θα πρέπει το μπαλάκι είναι στη δική σας πλευρά και θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό το οποίο μπορεί να βελτιώσει το κείμενο, αλλά είναι, εν πάση περιπτώσει, μια σύμβαση που έχει νομική βαρύτητα και βεβαίω η παραγωγή πρέπει να το έχουν αυτό για να μπορούν να έχουν ένα διάλογο και συνεργασία παρετέρω. Τώρα όσον αφορά ε, στην αλυσίδα όλη αυτή ο μετασχηματισμός που γίνεται νομίζω πως ελέγχθη προηγουμένως αλλά θα πρέπει να σας το πω με τον Επίτροπο Ταλιάνη με τον οποίο συνεργαζόμαστε και ο οποίος έχει σχέση με αυτό το φόρουμ το μεγάλο το οποίο συμμετέχουν και άλλοι επίτροποι με τα ε, γεωργικά και τρόφιμα για τα μέτρα κοινά τα οποία πρέπει να ληφθούν, ούτω ώστε ο ένα εργαζόμενος στη δικό του τομέα να φτάσουμε σε κοινέ θέσει όσον αφορά όλη αυτή την αλυσίδα των τροφίμων. Για το Γάλλο όμω ειδικά πιστεύουμε ότι το μίνιμουμ της διαφάνειας ε, το οποίο πρέπει να υπάρχει, πρέπει να εκτεθεί μέσα σε αυτό το κείμενο. Τώρα, σαν αφορά τη καταστάσεως της αγοράς, μπορώ, θα ήταν πολύ καλό να σας αποστείλω το κείμενο αυτή την ανάλυση την οποία έχουμε και αυτό το οποίο προς το παρόν μπορώ να σας πω είναι ότι οι αναλύσεις τις οποίες κατορθώσαμε να κάνουμε και οι οικονομικές αναλύσεις, η παραγωγή, παραγωγή θα είναι μικρότερη ε, καλύτερη διότι είναι πολύ αισιόδοξα για το 11 τα πράγματα και, πολύ, και βεβαίως υπάρχουν ε, καλύτερες οικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές άρα θα υπάρξουν αυτές με αυτές τις προοπτικές οι οποίες είναι ευνοϊκές με την προσθέμενη αξία με αύξηση της ε, κατανάλωσης των ε, τυριών και των γαλακτοκομικών προϊόντων και των φρέσκων, διαούρτια, κρέμες κλπ φαίνεται ότι θα αυξηθεί η παραγωγή κατά 8% από το 2009 ε, μέχρι το 2020 και τα τυριά επίσης κατά μισό της εκατό σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε. Αυτά όπως βλέπετε λοιπόν θα εξαρτηθούν όλα <clears throat> πώς το ευρώ θα εξελιχθεί καθότι εξαρτάται βεβαίω από την ευρωπαϊκή αγορά αλλά και από τη διεθνή αγορά, ιδιαίτερα για τα τυριά. Θα σα δώσω στόσο και να σας αποστείλω την ανάλυση εκεί η οποία χρειάζεται γραπτός για να βρείτε ελεπτομερή όλα τα στοιχεία αυτά. Όσον αφορά την καινοτομία τώρα, δεν προτείνεται σε αυτό το σημείο, καθότι το οποίο είναι κάτι το οποίο θα εξεταστεί στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής το 2013. Θα πρέπει να αλλάξουν όλα τα προβλήματα, τα εθνικά, τα τοπικά. Δεν ξέρω πραγματικά εάν με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε κερδίσει πολύ χρόνο. Εάν ανοίξουμε όλο το πακέτο το νομοθετικό όσον αφορά αυτό το θέμα μέχρι το 2014. Είναι κάτι βεβαίω το οποίο πρέπει να δούμε και το οποίο έχει σχέση με την καινοτομία και η καινοτομία ακριβώ θα πρέπει να ειδωθεί ιδιαιτέρως μέσα σε αυτά τα πλαίσια του όλου αυτού πακέτου θα λέγαμε μέχρι το 2014. Όσον αφορά την αναστάτωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή Ξέρετε, είχα επαφή με τη Γαλλική Προεδρία τους 20, ε, το οποίο προτείνει σε αυτό το σημείο να γίνονται οι μεταφορές οι οποίες γίνονται και οι συμφωνίες οι οποίες γίνονται, διότι είναι συμφωνίες αυτό ε, που έχει όσον αφορά το μετάβλητο αυτών των, αυτής της κατάστασης, ε, θα το υποβάλει η Γαλλική Προεδρία στο G20, στο G20 και εγώ το υπέβαλα επίση στο Προεδρείο κατά πόσον εξετάστηκε αυτό το πράγμα και για να ειδωθεί. Εάν το G20 είναι το καταλληλότερο φόρουμ για να θεθεί αυτό το θέμα. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες σε αυτό το θέμα είναι μέλη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτής της ομάδας η οποία θα δώσει τη γνώμη της και θα πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε αυτό το θέμα σε αυτό το επίπεδο που σας ανέφερα. Τώρα, όσον αφορά τους αριθμούς, πώς ακριβώς συμβόλαια υπάρχει, ο Λάιεν θέσατε ερώτημα με τις πολυεθνικές. Πιστεύω το ποσοστό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή και προτείναμε λαμβάνει υπόψη της, λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά τα πράγματα και νομίζω πως οι παραγωγοί έχουν αρκετή εξουσία, διότι οι πολυεθνικές έχει γαλακτοκομικά σε διάφορες περιοχές, σε διάφορα χώρες και συχνά εάν υπάρχει μια ελεξάρτηση μεταξύ των μεν και των δε και οι τιμές οι οποίες προτείνονται είναι διαφορετικές λόγω αυτής της διαφοράς που υπάρχει και το γάλα που διατίθεται διαφορετικά σε κάθε τοπική αγορά. Νομίζω πως αυτό το ποσοστό το οποίο προτείνεται μπορεί να συνάδει με αυτό το οποίο είπατε προηγουμένω, αλλά ο ανταγωνισμό στην αγορά σε εθνικό επίπεδο, διότι θα υπάρχουν πολλοί οργανισμοί οι οποίοι, τουλάχιστον τρει ή τέσσερι έχω πει ότι θα πρέπει να υπάρχουν, χωρί να υπολογίζονται μεταξύ αυτών των οργανισμών και οι συνεταιρισμοί οι οποίοι υπάρχουν και το γεγονό ότι υπάρχουν τέσσερι-πέντε, ε, συγκέντρωση τέσσερι-πέντε ανθρώπων στην, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο οργανώνεται αυτοί όλοι με τη μορφή συνεταιρισμών. Και οι συνεταιρισμοί συνεταιρισμοί έχουν μια ιδιαιτερότητα. Ότι δηλαδή η παραγωγή είναι εντό των συνεταιρισμών και εκεί γίνεται επεξεργασία. Έτσι λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο δεν μειώνεται η διαπραγματευτική αξία που έχει ο παραγωγός μέσα στα πλαίσια αυτών των συνεταιρισμών όταν έρχεται να διαπραγματευτεί. Αλλά αναλύσαμε τα πράγματα και όταν είδαμε τους αριθμούς αυτούς και είχαμε δεδομένα καθώς επίσης και μια δυνατότητα συσσόρευση, συσσόρευσης, μάζεψης αυτών όλων των στοιχείων ούτω ώστε ο παραγωγός φτάνοντας στη διαπραγμάτευση να γνωρίζει ακριβώς τα στοιχεία εκείνα τα οποία πρέπει να έχει κατά νου και να τα ολιγοπόλια σε εθνικό επίπεδο να μην λειτουργούν, γιατί υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί με τους συνεταιρισμούς, ξέρετε τι συμβαίνει, ε. σε 21 χώρες, εκ των 27, εκπροσωπούν πέρα των 20% οι συνεταιρισμοί και σε 17 είναι πέρα του 50% το γάλα που έρχεται από τους συνεταιρισμούς. Βλέπετε λοιπόν είναι ασχετά ισχυρή και ο κανονισμό, αυτό ο οποίο προβλέπει είναι να διατηρήσει αυτή την παραγωγή και 40%, 42% ε, είναι από τον άλλο τομέα το 42 και 58 σε όλο το ευρωπαϊκό επίπεδο έρχεται από του συνεταιρισμού, Το 58 επαναλαμβάνω. Συνεπώ. η Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου, η ΠΟΕ, ο τρόπος με τον οποίο προτείνει τη διαεπαγγελματική συνεργασία όπως λέγεται αυτή τη στιγμή για τον τομέα των ε, φρούτων και λαχανικών δεν νομίζω ότι πηγαίνει αντιτίθεται ε, αυτό που προτείνουμε εμείς με αυτό που προτείνει ο ΠΟΕ. Τα μονοπόλια σε ορευτικό επίπεδο δεν υπάρχουν, υπάρχουν συνεταιρισμοί δεν υπάρχουν συνεταιρισμοί στις νέες χώρες, στα νέα κρατημέλη. Νομίζω η Κύπρος, η Κύπρος αλλά δεν ξέρω ακριβώς, μπορεί η Κύπρος να έχει. Οι άλλες χώρες όμως έχουν, ε, οι συνεταιρισμοί έχουν πάνω από το 20% της αγοράς, οι παλιές χώρες θα λέγαμε. Ο κύριος Χάισιν μιλάει για την αλυσίδα των τροφίμων. Απάντησα λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί και να απαντηθεί, με βάση περιπτώσει θα πρέπει. Είναι ένα θέμα το οποίο θα εξεταστεί στα πλαίσια αυτού του πακέτου. Και συνεπώς ο κ. Φοντάνα για την παγκόσμια αγορά τι πρέπει να κάνουμε είπατε θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό μέσα σε αυτά τα πλαίσια του G20 του G20 όπως σας είπα και προηγουμένως αυτά Ευχαριστώ. Είχα μια προσανατολισμό. Ας αρχίσουμε με τα ερωτήματα των συναδέλφων. Ξέρετε, έχουμε πάρα πολλά γεγραμμένα να γνωρίζετε και θα πρέπει να δώσω καταρχήν και στο τέλος θα πρέπει να δώσω στον Επίτροπο ξανά το λόγο. Γι' αυτό θα σας παρακαλήσω να μένετε στο χρόνο σας με δύο λεπτά. Ο Γιώργος Παπαστάμκος πρώτος. Δύο λεπτά παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για την σταθερή δέσμευση για τη στήριξη του γεωργικού τομέα. Αναδείξατε κύριε Επίτροπε ορθώς ως κορυφαία προτεραιότητα την ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύω των παραγωγών έναντι των λοιπών κρίκων της διατροφικής αλυσίδας. Η εξισορρόπηση της διαπραγματευτικής θέσης προϋποθέτει την ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών. Με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα στηριχτεί η δημιουργία, η σύσταση και ο ρόλος των οργανώσεων παραγωγών. Επίσης, με ποια μέσα η παραγωγή θα είναι σε θέση να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά τους όρους των συμβολιακών σχέσεων, των contractual ε, relations, περιλαμβανομένης της τιμής με τους μεταποιητές γαλακτοκομικών προϊόντων. Και θα ήθελα κύριε Επίτροπε ε, να προσθέσω κάτι άλλο. Ε, σέβομαι πάρα πολύ, εκτιμώ πάρα πολύ αυτήν την ρυθμιστική σας την νομοθετική πρωτοβουλία για το γαλακτοκομικό τομέα. Όπως γνωρίζω τη σημασία του γαλακτοκομικού τομέα για ορισμένες χώρες, ε, αν θέλετε για τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Ε, επιτρέψτε μου να πω ότι ως Ευρωβουλευτής του Μεσογειακού Νότου και θα ήθελα αυτό να το ακούσει και ο κύριος Πρόεδρος ε, της Επιτροπής μας, θα ήθελα ε, να απευθύνω έκκληση για την ίδια. Δεν το λέω αντιθετικά, πολύ καλά κάνετε για τον ε, γαλακτοκομικό τομέα, αλλά για την ίδια ρυθμιστική εγρήγορση, για την ίδια κανονιστική ερύθμιση, εγρήγορση και για προϊόντα που έχουν τεράστια σημασία για τον Ευρωπαϊκό Νότο, όπως είναι το ελαιόλαδο, όπως είναι τα απορροκυπευτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Bravissimo Γιώργος, perfettamente in tempo. Σιεκερέσκι, c'ha la parola. Τέλεια, τηρήσατε το χρόνο, είσαστε συντομότατος κύριε Παπαστάμκο. Σιεκερέσκι, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα έπρεπε να αναλύσουμε τα βιώματα από τις χρηματοοικονομικές αγορές σε μεγάλο βαθμό έχουμε υπηρεσίες που υποτίθεται ότι εποπτεύουν τις αγορές. Εμείς όμως ακολουθούμε την αντίθετη κατεύθυνση. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες της γεωργικής παραγωγής και την κρίση το 2007, την επισητιστική κρίση, καθώς επίσης και την κρίση των γαλακτοκομικών στον τομέα αυτό το 2009, η παραγωγή γάλακτος έχει πολλές ιδιομορφίες ως ξεχωριστή παραγωγή και δεν είναι πολλοί οι οποίοι θέλουν να εμπλακούν και να παράγουν γάλα σε αυτόν τον τομέα. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα θέματα της συμπίκνωσης, επικέντρωσης, αν καταργηθούν ποσοστώσεις. Η παραγωγή θα επικεντρώνεται σε περιφέρειες που θα έχουν ευνοϊκούς όρους για τέτοιες παραγωγές και όπου θα υπάρχει και η σωστή υποδομή. Θα εξαφανιστούν οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις όταν θα βρίσκονται σε μειονεκτικές περιφέρειες. Θα συνεχίσουν όμως να παράγουν γάλα, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο σύστημα παραγωγής. Αν δεν, δεν υποστηριχθεί αυτή η παραγωγή θα εξαφανιστεί. Δεν θα υπάρχει πια ζωή σε αυτές τις περιοχές, σε αυτές τις περιφέρειες. Ένα άλλο πρόβλημα. Δεν κάνουμε συχνά λόγο για τις σχέσεις μεταξύ του μεταποιητικού τομέα για το γάλα και τις αλυσίδες διάθεσης των προϊόντων στις αγορές. Και αυτό είναι όμως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την επισητιστική αλυσίδα. Ένα άλλο θέμα. Έχουμε την ενιαία εσωτερική αγορά. Οι αποφάσεις όμως περιλαμβάνονται στις παγκόσμιες αγορές σήμερα. Πρέπει να αναλύσουμε λοιπόν την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και τι είδους προσέγγιση θα πρέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός ε, Εμπορίου να υιοθετήσει και πώς θα εμπλακεί. Έχετε εκπονήσει κάποια μελέτη επιπτώσεων για την πρόταση την οποία μας υποβάλλεται σήμερα. Πώς θα συνεισφέρει η πρότασή σας να υπάρξει σταθεροποίηση των πραγμάτων. Διότι μπορούμε να προβλέψουμε μια κατάσταση όπως και αγραφείτε ότι το 2014 θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ανάλυση των μέσων που έχουν καθελκιστεί και που εσείς παρουσιάζετε σήμερα και θα ληφθούν οι αποφάσεις αν θα διατηρηθούν οι ποσοστώσεις στα γαλακτοκομικά ή όχι. Και πολλά άλλα σημεία αξίζουν να αναφερθούν. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε τούτο. Ας δούμε τις ιδιομορφίες των γαλακτοκομικών προϊόντων και τις ιδιομορφίες της γεωργικής παραγωγής συνολικά. Ας μην ακολουθήσουμε την ατραπό που ακολούθησε ο προηγούμενος επίτροπος μιας πολύ, προς πολύ φιλελεύθερες λύσεις, διότι αυτό δεν είναι επωφελές για τη γεωργία και τους παραγωγούς. ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ εσάς κύριος Επίτροπε για το πακέτο για τα γαλακτοκομικά. Το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό μήνυμα έναντι των Ευρωπαίων παραγωγών σε αυτή την θα έλεγα οικονομικά πολύ τεταμένη περίοδο, κυρίως και για τα γαλακτοκομικά. Προσέξτε, είναι ένα, μια πολύ σημαντική και σωστή προσέγγιση όπως και στα ε, οποροκυπευτικά να ακολουθηθεί <coughs> μια παραλυτροχία και να υπάρξει ενίσχυση των ενώσεων παραγωγών. Με θετικό βλέμμα το αντιμετωπίζουμε ότι την ιδιομορφία και την κατάσταση των συνεταιρισμών σε αυτόν τον τομέα την αναγνωρίζετε και λαμβάνετε υπόψη στο πρώτο input στις προτάσεις σας για αυτή την κατάσταση και για την διαμόρφωση των τιμών. Ίσως αυτόν τον τομέα θα μπορούσατε να τον εξειδικεύσετε περισσότερο ή με άλλα λόγια το 2000 τα 2008 είδαμε ότι οι τιμές ε, ήταν καταρχήν υψηλές μετά είχαμε μερίδια αγορών που απολέστησαν όσον αφορά τα γαλακτοκομικά και οι τιμές στη συνέχεια και υπέστησαν τις ε, αρνητικές επιπτώσεις και μειώθηκαν πολύ σημαντικά. Ποιες ασφάλειες, διασφαλίσεις μπορούν να δοθούν όσον αφορά τους Ευρωπαίους παραγωγούς ε, στο μέλλον για να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Το θεωρώ πραγματικά αξιέπαινο και χαιρετίζω τις προτάσεις σας ε, στο παράδειγμα για τη διαφάνεια και για το παρατηρητήριο που θα δημιουργηθεί και θα λειτουργήσει ε, και θα υποπτεύει τις αγορές. Όμως ε, σε σχέση με αυτό το input, α, πολλοί συνάδελφοι το ανέφεραν, έχουμε το εμπόριο που δεν καλύπτεται, παραμένει εκτός ακόμα οι αλυσίδες και η διάθεση προϊόντων. Είχαμε την έκθεση του Ζωζέ Μποβέ που είχαμε εγκρίνει και που έχει πολλά συγκεκριμένα σημεία που εξειδικευμένα καταδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι το εμπόριο των ε, τροφίμων να συμπεριληφθεί, ιδιαίτερα όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σταθερό πλαίσιο τιμών για τους παραγωγούς. Τελευταία επισήμανση και απευθύνεται αυτή κυρίως σε εξειδικευμένες περιοχές με μειονεξίες, με μειονεκτικές περιοχές όπως ορεινές περιοχές. Το θεωρώ πολύ σημαντικό να υπάρξουν εξειδικευμένα μέτρα ώστε να υποστηριχθούν αυτές οι μειονεκτικές περιοχές στο μέλλον. Ευχαριστώ. Γκαρσία Πέρες παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Θα χρειαστούμε χρόνο για να μπορέσουμε να μελετήσουμε πιο νυφάλια και σε βάθος το περιεχόμενο αυτής της πρότασης. Στην παρέμβασή σας ε, θέσατε ερωτήματα. Ζητήματα που μπορεί να είναι ενδιαφέροντα. Δεν ξέρω όμως αν πραγματικά στην συγκεκριμενοποίηση αυτών των μέτρων θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε την σημερινή κατάσταση. Φαίνεται ότι αυτό το πακέτο είναι μια ανταπόκριση, μια απάντηση σε μια κρίση του γαλακτοκομικού τομέα. Υπάρχουν όμως άλλα προβλήματα και αληθεύει αυτό που είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα και πρέπει να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Θέλω να ξέρω σε αυτό το πακέτο μέτρων υπάρχει κάποιο μέσο πραγματικό που θα μπορέσει να διασφαλίσει ένα υπαρκές επίπεδο τιμών για να καλύπτεται η τιμή των παραγωγών για την παραγωγή αυτών των προϊόντων. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Πρέπει να κάνουμε λόγο όμως ε, για ένα επαρκές επίπεδο τιμών για να καλυφθεί η παραγωγή από πλευράς, ε, τα, ή τα έξοδα από πλευράς ε, των παραγωγών. Αναφέρθηκε από τον Επίτροπο η περιφερειακή ισορροπία. Κάνουμε λόγο για κατάργηση ποσοστώσεων το 2015 και εφ' εξής. Πώς θα είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την παραγωγή σε χώρες σαν τη δική μου, στην Ισπανία, όπου αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εγκαταλείψουμε ποσοστώσεις όπου είμαστε ελληματικοί. Αυτή τη στιγμή δηλαδή απορροφούμε πλεονάσματα από παραγωγές άλλων χωρών και όταν θα α, καταργηθούν αυτά τα, αυτές οι ποσοστώσεις, πώς θα είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε αυτές τις εκμεταλλεύσεις που είναι λιγότερο ανταγωνιστικές, που όμως διασφαλίζουν την ανάπτυξη της υπαίθρου, την σταθερότητα των περιφερειών και είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Μας απασχολεί και πρέπει να τεθεί αυτό το θέμα, να εξειδικευθούν μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ένα ζήτημα. Και αυτό είναι ότι σε αυτό τον τομέα, εφόσον ο παραγωγός φεύγει από την παραγωγή, αποχωρεί, δεν αντικαθίσταται από άλλους. Πρέπει να βρούμε μέτρα για την ισορροπία των πραγμάτων στις περιφέρειες. Να αναζητήσουμε την ανταγωνιστικότητα για εκείνες τις εκμεταλλεύσεις που βλέπουμε ότι πραγματικά πιέζονται ιδιαίτερα και αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστούμε. Η κυρία Πατράων Νέβες, δύο λεπτά. Μετά Γέκλε. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρίως για την παρουσία εδώ του κυρίου Επιτρόπου και πραγματικά για την παρουσίαση τέτοιων θεμελιωδών ε, εγγράφων μέσα από μια θέση διαλόγου και ε, προθυμίας ε, σημείωσα πολύ καλά αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και όπως και άλλοι συνάδελφοι δεν είχαμε και εμείς χρόνο να διαβάσουμε αυτό το έγγραφο. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν είναι μέτρα που είναι ουσιαστικά θετικά. Όμως επιτρέψτε μου κύριε Επίτροπε, κάνοντας λόγο εδώ κυρίως ως Πορτογαλίδα και από τις Αζόρες που προέρχομαι, να πω ότι αυτά τα μέτρα είναι ανεπαρκή, σαφώς ανεπαρκή για να καλυφθεί αυτός ο τομέας στη χώρα μου όπως πρέπει. Πρώτα απ' όλα και κύρια, επειδή δρά πάνω από την ε, ε, αλυσίδα αυτή. Έχουμε εμείς ε, σε σχέση με τους παραγωγούς και τη μεταπητική βιομηχανία ζητήματα. Ξέρουμε όμως ότι η γαλακτοκομική παραγωγή που έχει ε, υποστεί πλήγματα από κρίσεις και με τέτοιο ευμετάβλητο πλαίσιο τιμών πρέπει να τύχει ιδιαίτερη προσοχής. Όχι κατακαιρματισμένα αλλά ολιστικά, συνολικά που θα αντιμετωπίζει όλη την αλυσίδα και όχι μόνο το ένα σκέλος ή το άλλο. Και για την διαμόρφωση των τιμών. Ελπίζω ότι θα υποβάλλετε άλλες προτάσεις που θα έχετε εκπονήσει με άλλους επιτρόπους για να ληφθεί υπόψη αυτό το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή όμως είναι ανεπαρκή αυτά τα μέτρα για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Και όταν κάνουμε λόγο για καταστάσεις όπως στην Πορτογαλία, διαπιστώνουμε ότι εμείς στην Πορτογαλία έχουμε μία μόνη βιομηχανία που 70% έχει τις, παρα, την παραγωγής μας ε, και δεν ε, είναι εξαγωγική και όλα αυτά σημαίνουν ότι υπάρχει ένα μονοπόλιο de facto και όσο και ανεμένει και επιμένει κανείς στη διοργάνωση των ε, παραγωγών μέσα από τις ενώσεις τους δεν υπάρχει άλλος στον οποίο να μπορούν να πωλήσουν τα προϊόντα τους. Υπάρχει ολιγοπόλιο ή μονοπόλιο. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοιες βιομηχανίες και κάνετε λόγο για πολλές, διάφορες βιομηχανίες. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Δεν μπορούμε να σκοτώσουμε τον τομέα σε κάποιες χώρες και σε άλλες χώρες να ευδοκιμεί. Και τέλος για να ολοκληρώσω, ερωτώ, αν πραγματικά σε όσα αφορά, ολοκληρώνω, σε σχέση με την αξιολόγηση που κάνατε λόγο για αυτήν το 2014, αυτή η αξιολόγηση επιπτώσεων, αν αναγνωρίσει ότι είναι ανεπαρκής η χρήση αυτού του μέσου, όπως και για τις ποσοστώσεις, και εγώ πιστεύω ότι είναι ανεπαρκής, θα σκεφτούμε κάτι άλλο τη διατήρηση των ποσοστώσεων για κάποιο χρονικό διάστημα εφόσον δεν θα έχουμε επαρκείς μηχανισμούς για να διατηρηθεί σε λειτουργία σωστή η αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Γέκλε παρακαλώ. Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας χαρακτηρίζει ότι πολύ νωρίς αναζητείτε τον διάλογο μαζί μας και κανένας δεν μπορεί να αποκομίσει από εμά την εντύπωση ότι βρισκόσαστε πίσω από ένα τείχος ή τείχισμα και υποβάλλετε κάποιες προτάσεις σε ένα στεγανό πλαίσιο που δεν θα έχετε επαφή με την Επιτροπή Γεωργίας. Ή σας ευχαριστούμε που αναζητήσατε αυτή την επαφή μαζί σας. Ακούσατε πολλές παρατηρήσεις από εμάς και για μια πρώτη, α το πω έτσι, τοποθέτηση δώσατε και κάποιες απαντήσεις από πλευρά σας. Εγώ σας θεωρώ σύμμαχό μας

και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό να σκεφτούμε, να δούμε πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε. Ποια είναι τα επίπεδα στα οποία μπορούμε και πρέπει να σας υποστηρίξουμε και με ποιο τρόπο. Εγώ προέρχομαι από τη Νότια Γερμανία, από τα ελβετικά σύνορα, κοντά σε μια περιοχή κοντά στα ελβετικά σύνορα. Και το τι συμβαίνει στην Ελβετία καθημερινά και πολύ συχνά το παρατηρούμε στη συζήτηση αυτή. Είναι διασυνοριακά αυτά τα αποτελέσματα και στη Γερμανία θα έλεγα από την Ελβετία. Και δεδομένων αυτών πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά τι θα κάνουμε. Το θεωρώ πολύ σημαντικό ότι την ήπια προσγείωση, soft landing, θέλετε να το δημιουργήσετε, να το υλοποιήσετε και να αποκτήσει σάρκα και οστά. Είχαμε μια ανώμαλη προσγείωση μέχρι σήμερα και όχι ήπια και σε σχέση με την εξέλιξη των αγορών και των τιμών. Είναι σημαντικό σε τρία επίπεδα να δράσουμε. Το πρώτο επίπεδο είναι το πιο χαμηλό και επ' αυτού, το είπαν πολλοί συνάδελφοι, εντάσσονται σε αυτό το επίπεδο μειονεκτικές περιοχές και περιφέρειες που πρέπει με διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπιστούν από παραγωγές σε άλλες ε, περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλα χαρακτηριστικά. Επόμενο επίπεδο, η ενιαία εσωτερική αγορά και η διαφάνεια. Είπατε, σωστά, τα διεκδικούμε αυτά, διαφάνεια. Όμως όταν υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις πρέπει να υπάρχει κινητοποίηση και δράση. Μόνο να υποπτεύουμε και μόνο διαφάνεια δεν επαρκούν. Το επόμενο επίπεδο είναι το επίπεδο μέσα στο πλαίσιο της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μεταξύ των συναδέλφων σας επιτρόπων. Πιστεύω ότι πρέπει παντού όπου έχουμε τη δυνατότητα να καταστήσουμε σαφές ε, στους συναδέλφους σας επιτρόπους πού τα πράγματα πιέζουν και πού υπάρχουν προβλήματα. Θα πρέπει για την ενιαία εσωτερική αγορά να δράσουμε και να δούμε ότι βρισκόμαστε σε ανταγωνισμό παγκόσμια, σε παγκόσμια κλίμακα. Έρχομαι σε δύο σημεία. Είναι οι συμβάσεις, διμερείς συμβάσεις και συμβόλαια. Και οι συμβάσεις και συμβόλαια που συνάπτουμε με άλλες χώρες. Έχουμε και εκεί συμφέρον στα γεωργικά, τα συμφέροντά μα. Ε, να τα προασπίσουμε. Διεξάγεται ευρύτερη συζήτηση σε διαφορετικούς τομείς. Θα ήθελα σε εσά ως Επίτροπο, στο συνολικό σώμα των ε, Επιτρόπων, να υπενήσω αυτά τα πράγματα σε εσά και για τους κανόνες των χρηματοοικονομικών αγορών που συζητούμε να τους ε, μεταθέσουμε στο πλαίσιο αυτό των γαλακτοκομικών. Χρειαζόμαστε κανόνες. Ευχαριστώ. παρακαλώ, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα να επιστήσω την προσοχή σε ένα πράγμα που πολλές φορές γίνεται σαφές σε μένα στην δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Συζητάμε έντονα ποια προβλήματα υπάρχουν σε σχέση με γεωργούς και που δεν τα καταφέρνουν. Υπάρχουν όμως γεωργοί που εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες, προσαρμόστηκαν στις περιστάσεις και αντέδρασαν στην κρίση. Και αυτούς τους γεωργούς πρέπει να λάβουμε υπόψη σίγουρα. Και γι' αυτό αυτό το έγγραφο και υπό το δικό τους πρίσμα πρέπει να το εξετάσουμε. Να δούμε για αυτούς τους γεωργούς που ε, προσαρμόζονται στην αγορά και καταβάλουν προσπάθειες να μην υπερρυθμίσουμε τα πράγματα υπερβολικά και τους στραγγαλίσουμε. Και να δούμε και σε σχέση με όσους ε, δεν διαμαρτυρήθηκαν και δεν συμπορεύθηκαν με όσους ε, διαδήλωναν, να δούμε ότι ανέλαβαν το ρόλο της επιχειρηματικότητας, το επιχειρήν έδωσε λύσεις. Να δούμε λοιπόν σχέση με εκείνους που εργάζονται και βρίσκουν λύσεις, τι γίνεται έναντι των άλλων που δεν βρίσκουν λύσεις. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε αυτούς τους γεωργούς που προσαρμόζονται και είναι ανταγωνιστικοί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά την κρίση δεν ήταν μόνο οι γαλακτοπαραγωγοί που είχαν προβλήματα. Είχαμε και σε άλλες αγορές και αν στη δική μου περιφέρεια λάβω υπόψη τα όσα συνέβησαν έχουμε πάνω από διπλάσιους χείρο ε, κτηνοτρόφους που ασχολούνται με την εκτροφή χείρων από ότι σε σχέση με γαλακτοπαραγωγούς. Να μην τα αγνοούμε όλα αυτά. Παρακαλώ να ληφθούν αυτά υπόψη σε αυτό το έγγραφο. Να μην ξεκινήσουμε υπερβολικά σε αυστηρά πλαίσια, στενά πλαίσια για την υπερρύθμιση με μια τέτοια πρόταση. Πρέπει να προσέξουμε από τη μία ρύθμιση, να μην πέσουμε από τη μία παγίδα στην άλλη παγίδα υπερρύθμισης ε, και γραφειοκρατικής διαμόρφωσης των πραγμάτων. Είμαι γνώμων που έχουμε αυτό το έγγραφο Τώρα πρέπει σε βάθος να εξετάσουμε και να συζητήσουμε τι θα γίνει και στο τέλος να έχουμε κάτι που θα είναι πιο αηφόρο και με πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα για να μην πάνε τα πράγματα στραβά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε που τόσο γοργά και έγκαιρα μας δώσατε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για αυτό το έγγραφο. Κάποιες παρατηρήσεις υπό το δικό μου πρίσμα. Έρχομαι από την Ανατολική Γερμανία και αρχίσαμε στη δεκαετία του 90 όταν γίναμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαμε ποσοστώσεις, είχαμε αναφορά, ε, όγκους ή ποσότητες αναφοράς ε, ε, και έτσι λειτουργήσαμε. Δεν ήταν όμως ε, πλήρως διαχειρίσιμα αυτά τα στοιχεία των, ποσοτήτων αναφοράς. Πρέπει να υποστηριχθούν όλα τα μέτρα που ενισχύουν τη θέση των παραγωγών. Οι γεωργοί θα έχουν τη δυνατότητα πιο ενισχυμένα να διοργανώνονται και να μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις και συμβόλαια. Όταν λένε κάποιοι συνάδελφοι ότι αυτό ακόμα δεν είναι επαρκώς ε, ενισχυμένο και διοργανωμένο, ε, πρέπει να πούμε ότι όταν έχουμε έξι οργανώσεις ε, που μπορούν να ιδρυθούν ε, στη Γερμανία θα ήμουν χαρούμενος αν είχαμε έξι. Γιατί για παράδειγμα να υπάρχει προθυμία των ε, γεωργών και των παραγωγών να οργανωθούν σε αυτά τα πλαίσια. Δηλαδή εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή τη συνιστόσα. Θα πρέπει να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη θετική προοπτική και να διοργανωθούν οι παραγωγοί. Παρ' όλα αυτά, τα εξή σημεία θα έλεγα πρέπει να συζητήσουμε. Παρότι τίνουν περισσότερο και εντάσσονται στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, της κοινή αγροτικής πολιτικής. Παρ' όλα αυτά εντάσσονται και στον τομέα των γαλακτοκομικών. Χρειαζόμαστε, την, ε, ε, λαμβάνοντας υπόψη την εκπνοή των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, τη σταθερότητα ε, ενός πλαισίου. Το βλέπετε κι εσείς έτσι ότι χρειαζόμαστε μέτρα στήριξης των αγορών και σταθεροποίησής τους. Μετά, προγράμματα πράσινης ε, δράσης ε, θα πρέπει να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Τα πράσινα προγράμματα που είχαμε μέχρι σήμερα αφορούν την επέκταση παραγωγής και δεν είναι στη διάθεση των γαλακτοκομικών παραγωγών. Το βλέπετε κι εσείς έτσι επίτροπε ότι χρειάζεται το πρασίνισμα αυτών των παραγωγών να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα προγράμματα για αυτή την προοπτική, για αυτούς τους παραγωγούς. Συμφωνώ με την κυρία Γέκλε στο τρίτο. Τρίτο, πώς μπορούμε για τις... Ε, ε, έμεσες αυτές συμφωνίες, συμβατικές συμφωνίες να τις απαγορεύσουμε. Μπορούμε με το παρατηρητήριο να δράσουμε, να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε με το παρατηρητήριο εποπτεύοντας τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Σκοτά. Σκοτά. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο για την πρόταση την οποία κάνει. Η ομάδα υψηλού επίπεδου της Επιτροπής έχει κάνει μια καλή δουλειά και οι προτάσεις είναι σφαιρικά θα έλεγα ικανοποιητικές και αντικατοπτρίζουν τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Υπάρχουν όμως θέματα ακόμα. Ιδιαίτερα σχετικά με τον κανονισμό για τις συμβατικές σχέσεις. Υπογραμμίζεται εδώ ότι λόγω ακριβώς της ποικιλία που χαρακτηρίζει την εσωτερική αγορά δεν μπορεί να υπάρξει μια ενιαία απόλυτη ρύθμιση για όλες τις χώρες. Πρέπει παρόλα αυτά νομίζω να αποφασιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ελάχιστα επίπεδα διαπραγμάτευσης. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν μεμονωμένες συμφωνίες ανάμεσα στους παραγωγούς ατομικά και σε αυτά εργοστάσια στις επιχειρήσεις, αλλά ανάμεσα στις οργανώσεις των παραγωγών και τις επιχειρήσεις. Ελπίζω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμείνει επίσης και στην ανιχνευσιμότητα του γάλακτος εφόσον θέλουμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κρίση φανεί στο μέλλον στον τομέα αυτό με αποτελεσματικό τρόπο. Κλάες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, προσεγγίζω την πρότασή σας σαν μια κλιμακούμενη πρόταση βήμα προς βήμα για την διαμόρφωση των συνθήκων του γάλακτος στην αγορά. Είχαμε το όνειρο να έχουμε μια απελευθερωτική κίνηση και τώρα βλέπουμε ότι βήμα προς βήμα πρέπει να εργαστούμε οι στόχοι σας όπως διατυπώνονται χωρίς αμφιβολία είναι σωστοί. Για την πορεία πρέπει όμως να συζητήσουμε. Το έγγραφο δεν λέει τίποτα για την περιφερειακή ισορροπία. Σύντομα αναφέρθηκε αυτό πιο πριν και γι' αυτό η επισήμαση ότι το γάλα χρειάζεται συγκεκριμένη υποστήριξη για την έδρα των, γαλακτο, των γαλακτοπαραγωγών ανάλογα με τις περιφέρειες. Είσαστε υπέρ της ενίσχυσης ε, των παραγωγών στην αγορά. Δίνετε σαφή όρια. Λέτε να μην υπάρχουν μονοπόλια. Εντάξει, θέτω το ερώτημα, θα πρέπει νέες ενώσεις παραγωγών να συγκροτηθούν και να δημιουργηθούν διότι μέσα στο πρότυπο των συνεταιριστικών οργανώσεων ίσως αυτά δεν θα ταιριάξουν. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας γι' αυτό. Τι θα γίνει και ποιο καθεστώς θα έχουν οι συνεταιρισμοί γαλακτοπαραγωγών. Θα συνεργαστούν οι μεν με τους δε ή θα είναι σε αντιπαράθεση οι μεν με τους δε. Πρέπει να υπάρχουν οι σωστές υποδομές και όχι να τις υπονομεύσουμε και να τις καταστρέψουμε. Στη δική μου περιφέρεια όλοι οι γαλακτοπαραγωγοί είναι συνεταιρισμένοι. Με εκπλήσει που ακούω ότι οι άλλες περιοχές της Ευρώπης δεν ισχύει αυτό. Τελευταία ερώτηση. Ποια θα είναι τα ωφέλη από ένα τέτοιο ευρωπαϊκό ε, παρατηρητήριο που θα υποπτεύει τις αγορές. Σε μια πρώτη προσέγγιση βλέπω υπερβολικό γραφειοκρατικό βάρος και υπερβολικά περίπλοκο χαρακτήρα. Πείτε μας, ποια θα είναι τα ωφέλη που θα δώσει αυτή η πρόταση. Richard Hashword και μετά Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι με τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη δυνατότητα παρέμβασης στην αγορά ή, το ότι δεν υπάρχει λόγος για παρέμβαση σε κάποιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι οι αλλαγές σε επίπεδο ρυθμίσεων του ανταγωνισμού θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη βιομηχανία να αποκαταστήσει την ισορροπία της αγοράς. Θα ήθελα όμως να ζητήσω να είμαστε προσεκτικοί. Νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν ήταν αυτό το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο κλάδος Σχετικά με τη διαφάνεια, συμφωνώ ότι η ενημέρωση για τις αγορές είναι ένα καλό μέσο για να κινηθούν σωστά οι εμπλεκόμενοι στην αγορά αυτή. Μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, να βρούμε τρόπους σαν παράδειγμα ε, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και νομίζω ότι εδώ θα συμφωνήσω και με τον George Lyon όταν λέει ότι υπάρχει ανάγκη ίσως να υπάρξει ένας ombudsman σε κάθε κράτος μέλος έτσι ώστε να ελέγχεται η σωστή λειτουργία της αγοράς. Εκεί που απογοητεύτηκα όμως λιγάκι, γιατί δεν άκουσα κάτι το πιο θετικό σε επίπεδο προτάσεων, είναι γιατί θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει ε, τους παραγωγούς να ξεφύγουν από τη λογική της πρώτης ύλης. Η αδυναμία στη συγκεκριμένη περίπτωση ιδιαίτερα στον γαλακτοκομικό τομέα είναι πολλές φορές η εποχιακότητα της παραγωγής, ο εποχιακός χαρακτήρας. Και γι' αυτό θα ήθελα να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους να εξισορροπήσουμε τις αγορές αποτελεσματικότερα και έτσι θα προσθέσουμε αξία στις παραγωγές. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις προς την κατεύθυνση αυτή και νομίζω επίσης ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν και χρηματοδοτικά κίνητρα για τους συνεταιρισμούς να κάνουν έρευνες αγοράς για να βρουν τρόπους εξισορρόπησης της αγοράς αυτής και να προσθέσουν αξία μεγαλύτερη στα προϊόντα τους. Ευχαριστώ. Ντόρφμαν. Ευχαριστώ. Το γάλα δεν είναι οποιοδήποτε προϊόν της γεωργίας. Είναι ένα κέριο, κύρια σημασίας προϊόν της γεωργίας μας. Και γι' αυτό θα έλεγα, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με το γάλα. Θα έλεγα ότι σε πολλές περιφέρειες και περιοχές της Ευρώπης συμβαίνει αυτό και ιδιαίτερα έχω υπόψη τις δικές μου ε, περιφέρειες και περιοχές, ε, ορεινές ε, περιοχές και δεν υπάρχει εκεί άλλη εναλλακτική λύση για αυτές. Ή θα παράγει κανείς γάλα ή δεν υπάρχει άλλος, άλλη μορφή παραγωγής, γεωργικής παραγωγής. Και σίγουρα αληθεύει κύριε Επίτροπε, πρέπει να ενισχυθούν οι ενώσεις των παραγωγών. Όμως ιδιαίτερα για τις περιφέρειες και περιοχές για τις οποίες ανέφερα πιο πριν, τις ορεινές, η παραγωγή γάλακτος ήδη ρυθμίζεται μέσω συνεταιρισμών. Και εδώ σε σχέση με αυτό η πρότασή σας δεν δίνει τίποτα καινούριο και γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε κάποιες αυταπάτες ότι εκεί όπου το γάλα πωλείται σε μεταποιητικές βιομηχανίες. Ε, δεν υπάρχουν διοργανω... διοργανωμένες διαπραγματεύσεις τιμών. Είναι πραγματικότητα ήδη αυτό και πρέπει να λάβουμε υπόψη τέτοιου είδους πραγματικότητες ε, μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Θα έλεγα ότι πρέπει να μην είμαστε τίγρης χωρίς δόντια, αλλά να είμαστε αποτελεσματικοί, να μην παριστάνουμε τους τίγρης και να είμαστε αναποτελεσματικοί. Πρέπει να έχουν αποτελέσματα οι προτάσεις μας. Και όπως είπατε για τα ποροκυπευτικά, παράλληλη τροχιά, ναι, αλλά η διαφορά είναι ότι τα μέτρα εκεί οδήγησαν σε επιτυχία. Υπάρχουν λειτουργικά προγράμματα τα οποία έδωσαν καρπούς για τα ποροκυπευτικά. Και εδώ η προσέγγιση αυτή για το γάλα, αν δεν υπάρχουν κίνητρα που θα δοθούν, δεν θα πετύχουμε και να υπάρχει δυνατότητα χρηματοοικονομικά κίνητρα και ευνοϊκές, ευνοϊκή αντιμετώπιση για τους παραγωγούς να εισαχθεί. Διαφορετικά θα είμαστε αναποτελεσματικοί. Τίγρης χωρίς δόντια. Και εδώ προσθέτω τη φωνή μου σε σχέση με τις παρεμβάσεις για ποσοστώσεις που έγιναν πιο πριν. Έχουμε το παράδειγμα της Ελβετίας και θα έπρεπε να το εξετάσουμε σε βάθος το παράδειγμα και το πρότυπο της Ελβετίας και να δούμε τα λάθη που έγιναν εκεί να μην τα επαναλάβουμε εμείς εδώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ρόντους παρακαλώ. Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ Κυρίως χαίρομαι κύριε Επίτροπε που βρίσκεστε ανάμεσά μας σήμερα. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι είμαι απογοητευμένη ήμουνα απογοητευμένη όταν τα επτά σημεία της High Level Group, της ομάδας υψηλών, ε, ε, υψηλών βαθμών ε, υπαλλήλων μελέτησα. Και τώρα έχω απογοητευτεί και πρέπει να πω υπάρχει μεγάλη απογοήτευση σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα να τεκμηριώσω αυτά που λέω. Τέσσερα στοιχεία στο έγγραφό σας έχετε συμπεριλάβει. Πρώτον, οργανώσεις παραγωγών. Λέτε, στα κράτη-μέλη θα πρέπει σε σχέση με τις υποχρεωτικές ε, συμφωνίες και συμβάσεις ε, που θα ε, μπορούν να συνάπτονται τομεακά από οργανώσεις παραγωγών για να υπάρχει διαφάνεια. Για οργανώσεις παραγωγών μπορώ να σας πω στη Γερμανία μέσω του νομοθετήματος για τη δομή των αγορών, Mark Structure, τα έχουμε προσεγγίσει και δεν άλλαξαν τα πράγματα. Λέτε, 33% της παραγωγής σε εθνικό επίπεδο δεν μπορούμε να το υπερβούμε. Θυμάμαι ότι αρχικά είχαμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 75% ως στοιχείο. Θέτω το ερώτημα, τι γίνεται, επέβαλε τις απόψεις του ο Επίτροπος για τον ανταγωνισμό, έτσι. Και σε σχέση με αυτό, το 33% θα επαρκέσει για τις συμβάσεις και συμβόλαια. Μπορώ να σας πω για την σύναψη τέτοιων συμβολέων και συμβάσεων ήθιστε να γίνεται αυτό στη Γερμανία. 90%, 99% έχουμε τέτοιου είδους συμβάσεις στη Γερμανία. Αυτό όμως δεν επαρκεί για την διοργάνωση των παραγωγών τομεακά. Θα Προσβλέπω να δω ποιες επιπτώσεις θα έχει η πρόταση. Θα ωφελήσει ή όχι. Διαφάνεια. Το χαιρετίζω. Η διαφάνεια είναι είναι κάτι θετικό, τόσο το καλύτερο να την προαγάγουμε. Τώρα όμως έχουμε κυκλικές εξελίξεις στην αγορά, πάνω και κάτω της αγοράς, αυξήσεις, μειώσεις. Αν δεν εκπονήσουμε αποτελεσματικά μέτρα θα έχουμε και πάλι κυκλικά τέτοια σημαντικά προβλήματα. Δεν υπάρχουν για Γερμανούς πολλά νέα στοιχεία στο έγγραφό σας και τα προβλήματα τα είχαμε και εμείς στη Γερμανία ούτως ή άλλως. Δεν μπορώ να δω πώς θα μπορέσουν ενεργά να υποστηριχθούν οι παραγωγοί και να είναι ισότιμοι εταίροι έναντι των βιομηχανιών και των αλυσίδων εμπορίου. Ευχαριστώ. Grazie. Adesso Madame Lulling per due minuti e... Δύο λεπτά Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τώρα είδα και εγώ το έγγραφο αυτό σε μια γλώσσα την οποία καταλαβαίνω λίγο καλύτερα από τα αγγλικά τα οποία μου είχαν δώσει στην αρχή της συνεδρίας. Επιφυλάσσομαι λοιπόν να το αναλύσω πιο λεπτομερώς με μεγαλύτερη χρονική άνεση. Πάντως Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι εξέφασαν κάποιες ανησυχίες σχετικά με τα όρια τα οποία προτείνονται στο άρθρο 126. Θα ήθελα να μάθω πως τα όρια αυτά μπορούν να επηρεάσουν τις αγροτικές δομές, ιδιαίτερα σε κάποια μικρή χώρα, σαν τη δική μου. Στο Λουξεμβούργο το σύνολο της παραγωγής το οποίο αντιπροσωπεύει θα έλεγα το 0,1% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύνολο λοιπόν της παραγωγής αυτής γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας σε συνεταιρισμούς εκ των οποίων ο ένας συγκεντρώνει άνω του 60% του αριθμού των παραγωγών. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τα όρια αυτά του 33% πώς λειτουργούν, λειτουργούν σωρευτικά, αν κατάλαβα καλά. Ή στη συγκεκριμένη περίπτωση ο περιορισμός αυτός δεν αφορά τους συνεταιρισμούς των παραγωγών. Έχουμε έναν μεγάλο ε, τέτοιο συνεταιρισμό που αποτελεί ολιγοπόλιο στο Λουξεμβούργο, αλλά γύρω μας έχουμε την Τανόν, την Εστλέ, τη Γιοπλέ, τη Λουξλέ, η οποία συγκεντρώνει το 60% των παραγωγών βέβαια, 120 εκατομμύρια τόνους γάλακτος, αλλά παρόλα αυτά είναι μια μικρή επιχείρηση, η Λουξλέ, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διεκδικήσει αγορές σε επίπεδο τιμών. Δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τις προηγούμενες γαλακτοβιομηχανίες τις οποίες αναφέρθηκα σε επίπεδο τιμών. Μπορείτε λοιπόν κύριε Επίτροπε να με διαβεβαιώσετε ότι οι δομές αυτές ε, δεν εντάσσονται στα όρια σας, διότι αν πράγματι επιμένετε σε αυτό, τότε θα διαλύσετε δομές από την Λουξλέ. Ξέρετε ότι η Λουξλέ μάλιστα έχτισε πρόσφατα ένα, ε, ένα νέο, ε, μια νέα βιομηχανική μονάδα και αν δεν έχει τη δυνατότητα να την τροφοδοτήσει τότε θα πτωχεύσει και νομίζω ότι θα είσαστε υπεύθυνο ουσιαστικά για μια παραγωγική δομή ιδιαιτέρως αποδοτική σε επίπεδο ανταγωνιστικό. Ευχαριστώ. Καλινόσκι και κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να πω εδώ, Επίτροπε, υπάρχει ένα απόφημα σύμφωνα με το οποίο πρέπει να πούμε ότι το καλύτερο δεν είναι εχθρός του καλού. Και θα πρέπει έτσι να λάβουμε υπόψη στη συζήτηση αυτών των μέσων για τα οποία κάνουμε λόγο εδώ, για ε, τα μέσα τα οποία θα είναι χρήσιμα. Το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών του γαλακτοκομικού τομέα, αυτά, αυτό που θέλουν είναι μέσα, εργαλεία για να ρυθμιστεί η προσφορά του γάλακτος ε, σε αυτό που είναι η κατάσταση στην κοινοτική αγορά σήμερα. Να είναι κάτι παρόμοιο προς τις ποσοστώσεις. Κάτι που θα εγγυάται τα εισοδήματα αυτών των παραγωγών των γαλακτοκομικών σε αυτόν τον τομέα, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα ότι οι παραγωγοί δεν έχουν άλλες δυνατότητες δυνατότητες παραγωγής σήμερα. Μου λείπουν λεπτομέρειες και στοιχεία για αυτές τις συμφωνίες μεταξύ των δικτύων μεταποίησης ε, και των ενώσεων παραγωγών και όλα τα τμήματα, τους κρίκους της αλυσίδας. Αν εγκαταλείψουμε το σύστημα ποσοστώσεων, αυτό τι θα σημαίνει. Θα σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί με την αύξηση των μηχανισμών παρέμβασης που υφίστανται ή υφίσταντο μέχρι τότε. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, θα χρειαζόμαστε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση μεγαλύτερη υποστήριξη και παγίωση των πραγμάτων για να είμαστε ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά. Το ίδιο ισχύει και για τον γαλακτοκομικό τομέα, μέσα στο πλαίσιο του αντιμονοπολιακού αγώνα, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν οι παραγωγοί στον τομέα. Ε, κύριε Επίτροπε, έχουμε τελειώσει μόλις τις παρεμβαίνοντας και τώρα σας δίνουμε το λόγο για να απαντήσετε. Να κάνω ένα έτοιμο βέβαια και αναφέρουμε στο θέμα του προγράμματος για την παραγωγή. Ένα θέμα το Κοινοβούλιο ήθελε να το υιοθετήσει μέσα το ε, έκθεση την οποία έχει. Βέβαια είναι ιδιαίτερο θέμα να άπτεται του, του γάλακτος Πώ Πώς μπορούμε να το προστατεύσουμε και πώς αυτό το πράγμα να γίνεται καλύτερη προσφορά προς την αγορά. Μπορούμε επίσης να πάρουμε υπόψη μας αυτή την βούληση που εκέφερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή θα πρέπει να περιμένουμε το πακέτο για να το κάνουμε. Παρακαλώ, έχει το λόγο και απαντήστε σε ερωτήματα τα οποία σας ετέθησα. De le paquet Όσον αφορά το πακέτο ποιότητα, αυτό θα έρθει ως ούπο. Θα έρχεται και τους δύο κανονισμούς επί, επιτάπητος και εγώ με το μέρος σας βεβαίως. Θα, διε, θα καθησυχάσω την κυρία Λούλινγκ αμέσως. Η πρόταση δεν αφορά τους συνεταιρισμούς, το λέω σαφώς και περιφράστος. Οι συνεταιρισμοί και στη Δανία για παράδειγμα είναι 100% κάτω χώρο 90% άρα οι συνεταιρισμοί δεν θίγονται είναι οι παραγωγοί επεξεργάζονται το γάλα αυτό που προτείνουμε εμείς είναι, είναι σχέση με τους παραγωγούς μόνο τώρα εκείνους οι οποίοι δεν είναι συνεταιρισμού στο Λουξεμβούργο είναι λίγοι βεβαίω, αλλά αυτό ισχύει για μία χώρα, αλλά ισχύει και για το μέρος της αγοράς για τις υπόλοιπες χώρες δηλαδή μπορούν αυτοί να αποτελέσουν μέρος οργανισμών γειτονικών χωρών και άρα μπορούν να σωθούν θα το δείτε μέσα στον κανονισμό αυτό το πράγμα στο σχέδιο κανονισμού το οποίο έχουμε και ελεπτομερή υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία σας αναφέρω συνεπώς κύριε Ροντούς έλεγε ότι το συμβόλαιο δεν σαν την ε, γαλακτοκομική κρίση. Δεν έχω εγώ την πραγματική ότι η λύση αυτή η οποία θα λύσει όλα ως απομηχανής θεός. Υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί οι οποίοι μένουν, να γίνουν λαμβανωμένες της κρίσης επίσης για την αγορά και Όλα αυτά τα συμβόλαια δίνουν κάπου ή θα πρέπει να δώσουν ένα προσανατολισμό για μια σταθερότητα. Συμφωνώ μαζί σε αυτή η βεβαίωση, η σταθερότητα δεν μπορεί να είναι διαφορετική γιατί και η αγορά ανεβοκαταβαίνει. Ούτε μπορούμε να ξέρουμε πώ θα καταναλωθεί γάλα από του καταναλωτέ. Ωστόσο, αυτό που προτείνουμε δίνει μια ορισμένη προοπτική στην όλη υπόθεση μέσα στα πλαίσια αυτό το συμβουλίο και εφόσον βεβαίως έχουν την ποιότητα εκείνη και στον αριθμό αυτό του 3% τον οποίο αναφέρατε το είχατε προηγουμένω ότι εδώ μέσα σε αυτή την νόση ότι είπανε ότι α, υπάρχει πολλή γραφειοκρατία, πάρα πολλέ περιορισμοί και δυσκολίες. Ωστόσο ε, αυτό το οποίο κάνουμε επιτρέπει να υπάρχει ανταγωνισμό στην αγορά αλλά και οι παραγωγοί μπορεί να έχουν το βάρος εκείνο το οποίο χρειάζονται σε σχέση με, τα, με τους μεγάλους και εδώ μιλάω για την μικρή ε, παραγωγές και τις παραγωγικές μονάδες διότι ξέρετε τι θα κάνουν οι μικροί όταν βρεθούν επίση ενώπιον μια εταιρεία, αν θέλετε, ενό μεγάλου που αποθέτει το τρίτο τη χώρη χώρα θα αρκέσει για αυτού σε ένα μικρό ποσοστό το οποίο μπορεί να το διαπραγματευτεί με τη μεγάλη αυτή μονάδα την οποία υπάρχει. Αφενός είναι ο ανταγωνισμός αλλά αφετέρου υπάρχει δυνατότητα αυτή, το χαρτί το διαπραγματευτικό για να υπάρχει μια ισορροπία δυνάμεων όπου μπορούν να καθεστούν ίσοι μεταξύ τους οι δύο αυτοί οι παράγοντες. Ήδη άκουσα πολλά σχόλια τα οποία στοχεύουν και για το αναγνώρισε όσον αφορά την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Είναι κάτι το οποίο είχαμε πει πολλές φορές ότι θα πρέπει να υποστηρίσουμε τους παραγωγούς για να υπάρχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Αυτό το πακέτο το έχω πει δεν θα επιλύσει όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε ενώπιό μας υπάρχουν δομικά, υπάρχουν προβλήματα αγοράς, υπάρχουν προβλήματα καινοτομία, στήριξη σε ειδικέ περιοχέ και ούτε καθεξή. και αυτά όλα θα επανέλθουν στα πλαίσια τη αναθεώρηση τη ΚΑΠ. Βλέπετε υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να έρθουν και βεβαίω μερικά θέματα τα οποία ε, θα επανεξεταστούν πάλι και πολλά. Εδώ υπάρχουν ειδικά μέτρα τα οποία άπτονται αυτού και μόνο του θέματο το οποίο εξετάσουμε. Επίσης, η ενθάρρυνση όσον αφορά τη μεταρρύθμιση, πράγμα το οποίο έφερε ο κ. Επίσης, το ίδιο ισχύει όσον αφορά τις τοπικές βοήθειες οι οποίες πρέπει να γίνουν για την υποστήριξη, το αυτό ισχύει, ότι θα υπάρξει δηλαδή. Λαμπρά, τώρα, Όσον αφορά πολλές, ε, κύριε Ρέντινγκ, είπατε πολλοί κανονισμοί, πολλή γραφειοκρατία. Όχι, απλώ θα τα δίνουμε τη δυνατότητα στους παραγωγούς να οργανωθούν ε, δεν είναι υποχρεωμένο να το κάνει. Ο παραγωγό, ο οποίο βρήκε άλλη λύση, τόσο το καλύτερο για αυτόν. Όποιο ανήκει στο συνεταιρισμό, μπαίνει σε συνεταιρισμό και το καθεξή λαμπρά όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο θα του επιβάλλει αυτό τον κανονισμό. Αυτό ο κανονισμό θα έχει τα πλούστατα να προτείνει κανονισμού σε αυτού οι οποίοι έχουν προβλήματα, δεν είναι οργανωμένοι και του βοηθάει κατά αυτόν τον τρόπο να οργανωθούν κατά κάποιο τρόπο. Δεν νομίζω πω αυτό θα προτείνει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό το οποίο σα λέγω. Τώρα, όσον αφορά τη διαφάνεια, το είπα, όσον αφορά την αληθεία τροφίμων, δεν εξετάζεται εδώ μόνο, θα εξεταστεί πλήρως αλλού και θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι αφορά τα μέτρα και στην παρέμβαση που έχει κάνει για την περίοδο αυτή της κρίσης προτείνεται με την έκθεση η οποία είναι ε, συνημένη επί της αγοράς του γάλακτος σήμερα όπως έχει αυτή τη στιγμή και τα, οι ποσοστώσεις, οι διπλές ποσοστώσεις θα πρέπει να συμπαθυνήσω ότι η, κατάργηση των ποσοστώσεων είχε αποφασιστεί από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποφάσισε και το οποίο είχε νομοθετική ε, δοσηδικία τότε και το κατήργησε αυτό το πράγμα. Δεν είναι λοιπόν εμείς το οποίο το παίρνουμε σαν απόφαση. Ε, ακριβώς αυτό με την έκθεση η οποία έχει σχέση με, το, με την περίοδο μετά τις ποσοστώσεις θα δούμε κατά πόσα πραγματικά είτε εσείς είτε το Συμβούλιο δεν δεχθεί να υπάρχει μια ρήτρα όσον αφορά τη διαταραχή όπως λέγεται μια, η οποία θα επιτρέπει να ληφθούν μέτρα για να οθηθούν οι παραγωγοί για τη μείωση της παραγωγής τους μετά από αναλύσεις οι οποίες θα γίνουν της αγοράς και, της αγοράς και βεβαίως λόγω της πτώσης όλα αυτά της κατανάλωσης ενώ η παραγωγή παραμένει μεγάλη και αυξάνεται. Λοιπόν, αντί καλύτερα να παρεύουμε στην αγορά και να αποφύρουμε ορισμένα πράγματα και να πληρώσουμε εκ των υστέρων αυτή, ε, προς τα έξω, εμείς αντιμετωπίζουμε αυτή τη ρήτρα που σας ανέφερα η οποία θα επιτρέπει να υποστηρίξουμε και να προωθήσουμε τους παραγωγούς να μειώσουν την παραγωγή τους σε μια περίοδο περιορισμένη. Είναι μια ιδέα την οποία τη σκεπτόμαστε και την αναλύουμε αυτό το διάστημα. Donc, bon, je, Garcia Perez, Κυρία Γκάρσια είπε πρέπει να σας πω το για τα δομικά προβλήματα στο γάλα είναι θέματα τα οποία θα εξεταστούν ευρύτερα στα πλαίσια της αναθεώρησης της ΚΑΠ. Όσον αφορά τον καθορισμό τιμών, πώς θα γίνει αυτός. Και Κίστιγκερ μου το ρώτησε αυτό. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ των παραγωγών και αυτών που επεξεργάζονται το γάλα. Υπάρχει δεν ορίζουμε εμεί όλου του κανόνε οι οποίοι εισάγονται μέσα στη σύμβαση. Η σύμβαση είναι το συμβόλαιο ε, περιλαμβάνει πολλά μέρη αλλά στο σχέδιο αυτού του κανονισμού βάζουμε ορισμένα στοιχεία τα οποία θα είναι τα ελάχιστα τα οποία θα πρέπει να ισχύσουν για να έχει μια ισχύ το συμβόλαιο αυτό το οποίο γίνεται η σύμβαση που γίνεται μεταξύ των δύο μερών λαμπρά. Αυτά θα διαπραγματευτούν αυτές οι υποθέσεις, αυτά τα συμβόλαια. Όσον αφορά την ενίσχυση των οργανώσεων των παραγωγών, έλεγα προηγουμένω ότι στα πλαίσια του, δεύτερου πυλώνα θα υπάρχουν ε, μέσα εθαρρυντικά, τρόποι εθαρρυντικοί για μια οικονομική υποστήριξη όσον αφορά αυτό, ε, την στήριξη αυτών των οργανώσεων και όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία έχουμε το οποίο τους έχουμε αντιστοίχω για τα φρούτα και τα λαχανικά, άρα θα μπει και στο γάλα αυτό το πράγμα για να μπορούν πραγματικά να διαπραγματευτούν τη σύμβαση αυτή με τα γάλα τα οποία θέλουν και μπορούν βεβαίως να επενδύσουν όσον αφορά τη συλλογή του γάλακτο, την επεξεργασία του γάλα, τη μετατροπή του γάλακτος και όλα αυτά έχουν μια προστιθέμενη αξία. Όλο αυτό είναι ένα ξεκίνημα, ένα starter για τον παραγωγό και έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι στα πλαίσια αυτά θα έρθουμε με μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν την, τον παραγωγό. Προσπάθησα κυρίε και κύριοι να απαντήσω σε όλες και τις ερωτήσεις οι οποίες αιτήθησαν και βεβαίως υπάρχουν και ερωτάσεις, ερωτήσεις οι οποίες είχαν τις λεπτομέρειε όσον αφορά αυτό το πράγμα, τις οποίες δεν έχετε γραπτώσει. Νομίζω πως θα επανέλθω ε, ε, στην αρχή του επόμενου έτους να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Επίτροπε, ευχαριστώ λοιπόν τον Τάτσι Αντσιόλος. Η επόμενη συνάντηση τακτική της Επιτροπής μας είναι την 25η Ιανουαρίου. Αλλά θα τα ξαναπούμε μέχρι τώρα. Αν δεν σας δω στο Στρασβούργο, καλές γιορτές.